Good afternoon, ladies and gentlemen. Please take your seats. Καλησπέρα σας, παρακαλώ καθίστε. Είμαστε έτοιμοι. κηρύσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής ΡΕΤΖΙ Περιφερειακής Ανάπτυξης και θα ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Παρακαλώ, καθίστε. υπάρχουν ε, τροποποιήσεις, υποδείξεις για την ημερήσια διάταξη. Εάν όχι, θεωρώ ότι την εγκρίνουμε. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 16 και 17 Μαρτίου και 18 και 19 Απριλίου του 2016 αντιστοίχως. Το προσχέδιο πρακτικών είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Προτείνω, εκτός και αν έχετε αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της σημερινής μας συνεδρίασης, να θεωρήσουμε ότι εγκρίνουμε τα πρακτικά με το πέρας της σημερινής μας συνεδρίασης. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Έχω δύο να κάνω ανακοινώσεις. Έχετε αυτές τις κάρτες στο τραπέζι σας. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ε, αργία στη Βουλγαρία και στις σλαβικές χώρες. Σήμερα γιορτάζουμε το σλαβικό αλφάβητο. Είναι θέματα που άπτονται της κουλτούρας και του πολιτισμού μας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε παρακαλώ αυτό το κείμενο, λέει ο κύριος Φανίλ Στελρό, γιατί δεν ξέρω τι μου λέτε με αυτή την ε, κάρτα. Είναι το αλφάβητο, το δικό μας, το κυριλικό μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να προσπαθήσετε να γράψετε στα βουλγαρικά ή στα ρωσικά. 300 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίω χρησιμοποιούν αυτό το αλφάβητο. Μπορείτε και εσείς να μπείτε σε αυτή την κοινότητα ανθρώπων. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τη σημερινή μέρα η οποία είναι μέρα εθνικής εορτής ε, στη Βουλγαρία. Και με αυτή την ευκαιρία ε, εορτάζουμε τον πολιτισμό, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, ε, τον αλφαβητισμό ε, στις χώρες μας. Δεύτερο, δεύτερη ανακοίνωση. Αντιπροσωπεία στην Κροατία. Η Επιτροπή μας απέστειλε, οργάνωσε μια αποστολή στην Κροατία, όπως γνωρίζετε, και το πρόγραμμα περιλάμβανε συναντήσεις στο Ζάγκρεπ με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τον αρμόδιο Υπουργό και με το Εμπορικό Επιμελητήριο, με εκπροσώπους αυτού και στο συμπαίνει με τοπικές και περιφερειακές αρχές. Και η αποστολή μας επισκέφθηκε και έργα που έχουν ε, χρηματοδοτηθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία και αναμένεται να αποσταλεί έκθεση μέχρι τα τέλη αυτής της εβδομάδας. Ο κ. Κοτσολίνο ήταν επικεφαλής της αποστολής ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ρέτζη και θα ήθελα να του δώσω το λόγο για να μας πει δύο λόγια για την αντιπροσωπεία. Ωστόσο δεν βρίσκεται μαζί μας. Τα άλλα μέλη της αποστολής ήταν ο κύριος Φανίστερο και ο κύριος Νοβάκοφ, η κυρία Μάλετιτς και η κυρία Τόμασιτς, αν δεν απατώμε. Ε, θέλει κάποιος να πει κάτι. Παρακαλώ κύριε Φανίστελ Ναι, εν συντομία. Κυρία Πρόεδρε, για αυτή την αποστολή της αντιπροσωπείας μας. Αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι η, η χώρα έκανε εξαιρετική δουλειά. Κατάφερε να ενώσει όλο το έργο της πριν από την προσχώρησή της με τη δουλειά που ξεκίνησε άπαξ και προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι μπόρεσαν να αξιοποιήσουν όσο δυνατόν περισσότερα κονδύλια και να επιταχύνουν το ρυθμό των εξελίξεων. Υπάρχει μεγάλη ελπίδα και ότι η οργάνωση και η διοίκηση είναι σε θέση να επιτελέσει αυτό το έργο τα μέσα μαζικής επικοινωνίας αναμεταδίδουν το έργο αυτό και η σημερινή κυβέρνηση έχει επιφέρει κάποιες αλλαγές σε, προγραμματικό επίπεδο ως προς την αξιοποίηση των κονδυλίων, ε... συνάπτει συμφωνίες με εταιρικές σχέσεις, ε, συνάπτει συμφωνίε με νέου εταίρου και δημιουργεί νέε εταιρικέ σχέσει. αυτό βέβαια υπάρχει, ε, δημιουργεί κάποια χρονικά κενά, γιατί οι νέε συμφωνίε πρέπει να περάσουν από το Κοινοβούλιο, επομένω κάποια βρίσκονται, ε, γίνονται σε κενό χρόνο. Το reprogram είναι ο επαναπρογραμματισμός, είναι μια πολύ εύυχη λέξη, ωστόσο ο υπερβολικός επαναπρογραμματισμός μπορεί να οδηγήσει σε πολλές αβεβαιότητες. Αυτό καταρχάς ήταν ένα πρώτο συμπέρασμα και μια πρώτη διαπίστωση. Δεύτερον, η δυνατότητα των περιφερειών να δουλέψουν οι εκπρόσωποι των περιφερειών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πόλεων, των δήμων δηλαδή, ε, μας μίλησαν για το κύριο μέλημά τους που είναι να διατηρήσουν το στελεχειακό τους δυναμικό. Ε, ε, άξια στελέχη, άξιους ανθρώπους νέους να μείνουν ε, πρώτα στη διοίκηση, ωστόσο μετά δυσκολεύονται να τους κρατήσουν γιατί το θεωρούν ως εφαλτήριο για να μεταπηδήσουν στον ιδιωτικό τομέα όπου οι αμοιβέ θα είναι υψηλότερες. Ξέρετε, είναι δύσκολο για εμάς από τις κάτω χώρες όπου έχουμε πολύ υψηλότερους μισθούς Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν για χρόνια ολόκληρα στην εκάστοτε διαχειριστική αρχή και η δουλειά στη διαχειριστική αρχή λειτουργεί ως εμφαλτήριο για άνοδο, για επαγγελματική ανέλυξη, για ε, ενίσχυση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Και αυτό καταρχάς δηλαδή ότι υπάρχει κίνδυνος ότι έρχονται στελέχοι, μαθαίνουν και μετά μπορεί να τα χάσουν γιατί μεταπηδούν στον ιδιωτικό τομέα. Από εκεί και πέρα πήγαμε και στις πόλεις και είδαμε ότι κάποιες πόλεις κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και αξιοποιούν τα κονδύλια, ενώ ε, στα ε, χωριά στην Ήπεθρο πραγματικά υπάρχει έλλειψη. Προσπαθούν να παρέχουν υπηρεσίες για νέους, για παιδιά, για ηλικιωμένους. Στρέφονται ο κόσμος της Ήπεθρου με τα μάτια ορθάνυχτα προς την Ευρώπη δεν ήταν τόσο περίπλοκοι οι κανόνες πριν από την προσχώρηση της χώρας αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους δυσκολεύει το περίπλοκο νομικό πλαίσιο τους δυσκολεύει το ότι πρέπει να εκπληρώσουν διάφορα κριτήρια που είναι αναγκαιότητα. Καλό είναι λοιπόν να ξανασκεφτούμε και εμείς τι είναι αυτό που κάνουμε. Τρία είναι τα βασικά μηνύματα κάνετε πολύ επαναπρογραμματισμό στο μέσο της διαδρομής. Δεύτερον, σκεφτείτε αν έχετε πραγματικά τους ανθρώπους στα διάφορα επίπεδα της διοίκησης που χρειάζεται. Και τρίτον, η πολιτική σας, εάν πραγματικά καλύπτει τις ανάγκες ε, της υπαίθρου, του κόσμου που ζει στην υπαίθρο. Σε κάθε περίπτωση ήταν πάρα πολύ καλές οι συναντήσεις μας. Και τα μέλη του Κοινοβουλίου έπρεπε πάντοτε να είναι υπατμόν. Το πρόγραμμα ήταν πολύ βεβαρημένο, οι οδηγοί το πολύ να περίμεναν μισή ώρα κάπου. Είχαμε πολλές και διαφορετικές εμπειρίες, δηλαδή καταφέραμε να συλλέξουμε. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά, όλους όσοι δούλεψαν για αυτή την αποστολή και μας βοήθησαν στις δύσκολες στιγμές. Ευχαριστούμε. Έχουμε εδώ και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Σαντρίν Τεμπουγγενό. Θα θέλατε να πείτε και εσείς δύο λόγια. Yes, good afternoon. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που επισκεφθήκατε την Κροατία. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, συνεισφορά σας. Είναι μια χώρα που έχει επενδύσει πολύ για να υποφελθεί όσο το περισσότερο από τα ταμεία μας και από τους πόρους μας. Βέβαια βρίσκονται σε μια καμπύλη εκμάθηση αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζουν πολλές ε, δυσκολίες αυτής της ε, πρώιμης ηλικία και μία από αυτές είναι η δυνατότητα να προσελκύσουν ε, και να διατηρήσουν αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή τη στιγμή συζητάμε μαζί τους τι είδου μέτρα στην πράξη θα μπορούσαν να πάρουν έτσι ώστε να διευκολύνουν ε, αυτή την διαδικασία της στρατολόγησης και της πρόσληψης ε, ανθρώπων αξιόλογων που θα αμείβονται βέβαια ανάλογα και με την ε, επίδοσή τους και προφανώς ειδικευμένους σε κάθε τομέα. Επίσης προσπαθούμε να τους επίσουμε να εξυγχρονίσουν το σύστημά τους, να το απλοποιήσουν γιατί και εμείς οι ίδιοι έχουμε διαπιστώσει το πόσο βαρύ είναι το σύστημα, το πόσο δυσκίνητο ε, πρέπει να είναι πιο ευέλικτη έτσι ώστε να είναι και πιο αποτελεσματική. Επίσης ε, προσπαθούμε οι διαχειριστικές ε, αρχές να γίνουν αυτόνομες και να έχουν μια αυτόνομη ικανότητα διαχείρισης των έργων. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι στα πρώτα τους βήματα, πρέπει να αναπτυχθούν δεν είναι απλό, διότι αυτή τη στιγμή ε, δεν έχουν ε, ένα μεγάλο αριθμό όριμων έργων. Οπότε θα πρέπει να δημιουργήσουν έτσι ένα pipeline από ε, έργα, όριμα έργα και ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικοί, να αναπτύξουν τις ικανότητες λήψης αποφάσεων και διαχείρισης έργων. Το παίρνουν πολύ στα σοβαρά αυτή τη στιγμή ορίζουν, ε, επεξεργάζονται το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης γιατί καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται να βοηθήσουν τον εαυτό τους να υποφεληθούν ακόμα περισσότερο. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να εργάζεται κανείς μαζί τους. Το δουλεύουν. Thank you. Thank you very much. We the Ευχαριστώ πολύ. Θα περιμένουμε την έκθεση που θα ετοιμάσει η Γραμματεία και θα μας ε, στείλει, θα στείλει σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, περνάμε στις ε, ψηφοφορίες. Καταρχήν θα ψηφίσουμε την ε, ε, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα ε, γνωμοδότηση πρωτοβουλία, η συγγήτρια είμαι εγώ ίδια. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο, πρώτη συμβαστική πρόταση. Είμαστε έτοιμοι. Συμβαστική πρόταση υπάρχει μόνο ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση υπαρθμών 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση υπαρθμών 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ. Τροπολογία 35 λέω υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση παριθμών 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 7. Όχι. 6. Διορθώνει η πρόεδρος. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 ε, συμβαστική πρόταση 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 69 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τρο... Συμβαστική πρόταση 10 υπέρ. Κατά. Ποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση παρθυμών 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρόταση 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 136. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 143 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 25 υπέρ. Κατά. εποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 148 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ κατά εποχές ε, εγκρίνεται. 150 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 26 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 27 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 166 Επέρ κατά ηλεκτρονική επιβεβαίωση για την τροπολογία 166 Άρχιτη ψηφοφορία The vote is closed. Λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται τροπολογία 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 ε, Σημαντική πρόταση 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω αλλά στο ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση, ε, συγγνώμη, τροπολογία 176. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 179. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 180 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι αναφορές πρώτη αναφορά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, εκτιμώντας τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές Ας το ελέγξουμε. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές. Ας το ελέγξουμε. Τροπολογία 12. Ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. The is closed. Λίγη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 και 14 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση. Α, πρέπει να ψηφίσουμε τη 15. Ποιο είναι υπέρ τη 15. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται. The vote is closed. Λίγη. Ε, έχουμε μία παραπάνω ψήφους από το ΕΛΚ. Πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Λυπάμαι. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη, αλλά η, ψήφος πρέπει να, η ψηφοφορία πρέπει να επαναληφθεί. Επαναλαμβάνουμε την τελική ψηφοφορία. Άρχεται. The vote is closed. Λίγη. Εγκρίνεται η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. We continue now with the opinion preparation of the Συνεχίζουμε λοιπόν με την ε, προετοιμασία του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 ε, πρόταση του Κοινοβουλίου ε, πριν από την πρόταση Κομισιόν. Κυρία Κρέλ, η συγγήτρια, θέλετε να πείτε κάτι. Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα δηλαδή ξεκινάμε με την ψηφοφορία. Και ξεκινάμε με την συμβαστική πρόταση ΠΕΡΤΜΟΝΕΝΑ, 1. Υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρόταση 2. Υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. τροπολογίες 11 και 12 καλύπτονται από το συμβαστικό κείμενο. Εγώ αυτό το κείμενο ψηφοφορίας έχω μπροστά μου. Τι να σας πω, λυπάμαι. Λοιπόν, είχαμε σταματήσει τη συμβαστική 3 που είχε εγκριθεί. Πάμε τώρα στη συμβαστική 4. Εδώ έχουμε ψηφοφορία σε τμήματα. <clears throat> σε δύο τμήματα για την 4. Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα τη 4. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. Η 53 παρακαλώ, για την 53 υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρι... Ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 8 και πάλι ψηφίζουμε σε τμήματα, σε δύο τμήματα, το πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Μισό λεπτό. Στο δικό μας τον ε, κατάλογο ψηφοφορίας, ε, τουλάχιστον ε, των μερών του ΕΛΚ, εδώ έχουμε την έκθεση ΚΡΕΛ, αλλά εγώ παρακολουθώ την έκθεση μιας άλλης έκθεσης. Να προσέξετε οι υπόλοιποι, να πάτε στην τελευταία έκθεση, εκεί να ψηφίζετε για την τελευταία, όχι για άλλη έκθεση. Ωραία λοιπόν. Πάμε στο δεύτερο τμήμα της 8. Ε, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. Η 64 παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 9 σε τμήματα, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 73 υπέρ, κατά, αποχές ε, νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Για την 73 ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε η γνωμοδότηση. Συγχαρητήρια. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε τώρα με την ε, γνωμοδότηση του κυρίου Νοβάκοφ ε, πώς μπορεί κανείς ε, να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο το δυναμικό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κύριε Νοβάκοφ, θέλετε να πείτε κάτι? Όχι. Πολύ ωραία. Κατόπιν τούτου περνάμε τώρα στην ε, ψηφοφορία και ξεκινάμε με τη συμβαστική 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 10, ε, ε, τροπολογία 10, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Για την 11, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, ε, πρέπει να προβούμε σε ηλεκτρονική επαλήθευση. Για την 11 παρακαλώ, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 16 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίφθηκε η 16. Αλλά ας ε, κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Για 16 ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Λυπάμαι, λυπάμαι, είχα κάνει λάθος. Συμβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 29, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. γιατί δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 29. Παρακαλώ, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίθηκε. 30. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίθηκε η συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 41 παρακαλώ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Η τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Θέλετε επαλήτευση. Λοιπόν, ε, ελέγχος ηλεκτρονική επαλήθευση για την 52, παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίθηκε. Η 54. Ε, υπέρ παρακαλώ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Η 55. Υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Οι 56 και οι 57 ε, ταυτόσημες ψηφίζουμε από κοινού και για τις δύο υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η 59 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 60 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 62 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσαμε για την 44, την τροπολογία. Ε, για τη 44 δεν ψηφίσαμε. Διότι εγκρίναμε την 29. Πολύ ωραία. Λοιπόν, περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε η γνωμοδότηση συγχαρητήρια. Και προχωράμε πρόσβαση ε, στη χρηματοδότηση από πλευράς μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ε, διαφοροποίηση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μια αγορά, ε, σε μια στην κεφαλαγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συγητής δεν θέλει να πει τίποτα. Ξεκινάμε λοιπόν με τη συμβαστική 1, υπέρ παρακαλώ, κατά ποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 11 υπέρ, κατά, αποχές ε, πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. 11 ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίθηκε. Η 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Η 28 προφορική τροπολογία. Ε, υπάρχει κανείς που να διαφωνεί, από ό,τι βλέπω όχι, πολύ ωραία. Άρα ε, Ψηφίζουμε για την 28. Ε, υπέρ παρακαλώ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Ε, υπέρ παρακαλώ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 58, προφορική τροπολογία. Ε, δεν ξέρω αν διαφωνεί κανείς με αυτή την προφορική τροπολογία. Για την 58 ψηφίζουμε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Η 77 παρακαλώ υπέρκατα κατά αποχές εγκρίνεται η 80 υπέρ κατά αποχές ε, ας ε, κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την 77 ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίζουμε παρακαλώ όχι για την 80 συγγνώμη έκανα λάθος τροπολογία υπερθμών 80 Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η 7. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Η τροπολογία 71. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και πάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. The vote Έκλεισε η ψηφοφορία. Και η γνωμοδότηση εγκρίθηκε συγχαρητήρια. Και κλείσαμε και με τις ε, ψηφοφορίες. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη α, είναι η συνάντηση με τον κύριο Κατάινεν που θα έρθει στις 4. Ε, Έχει έρθει. Ζητώ συγγνώμη. Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων.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 Okay, Ωραία, περνάμε στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξη. Ανταλλαγή απόψεων για το Ταμείο Ελληνικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιολόγηση. Συγητής ο κ. Τσίκο. Είναι μαζί μας και έτοιμος, πανέτοιμος να μας παρουσιάσει τις απόψεις του για την έκθεση. Παρακαλώ. Ε, σας παρακαλούμε το μικρόφωνο του ομιλητή, είναι κλειστό, δεν ακούμε. Σέντε. Sente? Il Fondo di solidarietà dell'Unione Europea Λοιπόν, κοιτάξτε, το Ταμείο Λεγγύης συστήθηκε το 2002 και όπως πολύ καλά γνωρίζουμε δεν μπορούμε να προβλέψουμε ε, όλες τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όμως μπορούμε να προσπαθήσουμε να αγγιηθούμε ε, να είναι πιο σωστή η αντιμετώπιση των ε, συνεπειών. Γνωρίζουμε λοιπόν όλοι ότι μια φυσική καταστροφή περνάει από διάφορες φάσεις. Η πρώτη φάση είναι το ότι ανακαλύπτει κανείς ότι είναι αδύναμος μπροστά στη φύση, ότι ότι δυστυχώς δεν μπορούσε να προβλέψει. Προσφέρεται άμεσα βοήθεια μέσα από τις υπηρεσίες διάσωσης, τις εθνικές και τις ε, διεθνείς και αυτή είναι η επόμενη φάση. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι ακριβώς αυτό, γιατί από τη στιγμή που ε, υπάρχει άμεση βοήθεια, ε, τα θύματα στην επόμενη φάση θέλουν την αποκατάσταση των ζημιών. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι θα πρέπει στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καταστήσουμε σαφές ότι η Κομισιόν οφείλει να λάβει υπόψη στο γεγονός ότι τα θύματα πολλές φορές δικαιολογημένα αισθάνονται εγκαταλελειμμένα. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να αξιολογηθούν όλες οι φάσεις. Το 2014 είχαμε τον κανονισμό για το Ταμείο Αλληλεγγύης. Τροποποιήθηκε αυτό για να υπάρχει καλύτερη λειτουργία του Ταμείου αλληλεγγύη. Θέλω να σας πω ότι βεβαίως και υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις από τον κανονισμό. Παραδείγματο χάρη να επεκτάθηκε το χρονικά διάστημα για να μπορεί κανείς να ζητήσει αποκατάσταση για φυσική καταστροφή από 12 σε 14 εβδομάδες. Επίσης περιορίστηκε ο χρόνος για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μέσα σε 8 εβδομάδες πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση και η Επιτροπή οφείλει να αποφασίσει ε, στο ελάχιστο χρονικό διάστημα. Επίσης προβλέπεται και δυνατότητα προκαταβολής του 10% της βοήθειας που θα χορηγηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα η Επιτροπή των Περιφερειών καλείται να αξιολογήσει την έκθεση που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το Ταμείο Λεγγύης και τα σχετικά κονδύλια τα οποία εκταμιεύτηκαν το 2014. Η ίδια Επιτροπή, αυτή η δική μας, πήρε 13 ε, ερωτήσεις για παροχή βοήθειας. Από αυτές οι 7 έγιναν δεκτές, οι δύο απορρίφθηκαν και οι υπόλοιπε ε, μεταφέρθηκαν στο 2015. Έτσι λοιπόν το 2014 126 εκατομμύρια ευρώ εγκρίναμε στο πλαίσιο ή με τη μορφή των κονδυλίων αλληλεγγύης. Ε, μας εστάλει λοιπόν η Επιτροπή η έκθεση από την Επιτροπή και είχαμε τις επαφές μας με τις ε, τοπικές ε, αρχές. Ε, θα πω απλά το τι σκεφτήκαμε. Ο μηχανισμός αυτός είναι ένα εργαλείο απολύτως απαραίτητο για να μπορούμε να αντιδράσουμε σε περίπτωση μεγάλης καταστροφής που λαμβάνει η χώρα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη χρηματοδότηση όλων των διαδικασιών προσπαθούμε να επαναφέρουμε την υποδομή, παραδείγματο χάρη, παροχή ηλεκτρικού ρεύματο, ε, νερού, ε, τι ε, απαραίτητε εκείνε ενέργειε που πρέπει να λάβουν χώρα για να μπορούν να ικανοποιηθούν οι άμεσες ανάγκε. Πρέπει να τεθούν σε ισχύ όλα τα μέτρα που αφορούν και στην προστασία της εθνικής κληρονομιάς. Οι θεομηνείς, οι φυσικές καταστροφές στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Σλοβενία ε, κατά τραγικό βαθμό ε, έπληξαν τις περιοχές. Στη δική μου την περιοχή, στην Σαρδινία, το 2013 είχαμε 16 θανάτους ε, και πάνω από 700 εκτοπιστέντες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις στήσεις τους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ήταν μεγάλη οικονομική ζημιά, το οποίο έτυξε τους ε, πολίτες. Και ε, πρέπει να πούμε επίσης ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι φυσικές καταστροφές έχουν πλήξει κυρίως τη Νότια Ευρώπη, που έτσι και αλλιώ έχουν πληγεί από την παγκόσμια κρίση. Με βάση τον κανονισμό του 2014, όπω σα είπα, ε, περιορίζεται ο χρόνο εκταμείευση των κονδυλίων. Πρέπει να γίνει μέσα σε έξι εβδομάδε από τη στιγμή που γίνεται δεκτή η αίτηση. Εγώ πιστεύω ότι ο χρόνο που είναι απαραίτητο για να κινητοποιηθούν τα κονδύλια ακόμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άρα δηλαδή θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρώτα απ' όλα να εστιάσει την προσοχή του στο τι είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα των διοικητικών διαδικασιών που προβλέπονται για την κινητοποίηση του ίδιου του Ταμείου. Για την αλήθεια ότι μιλάμε για έξι εβδομάδες, αλλά για να σας κάνω πάλι ένα παράδειγμα από τη Σαρδινία, την πατρίδα μου, ε, το 2013 η Σαρδινία θα έπρεπε, ήταν αναγκασμένη να περιμένει 1,5 χρόνο για να πάρει τα κονδύλια από τον Νοέμβριο του 2013 που κατετέθη το αίτημα. Τελικά τα κονδύλια έφτασαν το 2015. Άρα δηλαδή μιλάμε για ένα χρόνο αντικειμενικά πάρα πολύ μεγάλο. ω εκ τούτου οι πολίτε αισθανόντουσαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα εγκαταλελειμμένοι. Είναι λοιπόν απαραίτητο να βελτιωθούν οι γραφειοκρατικέ διαδικασίε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να περιοριστεί το χρονικό διάστημα, όπω σα είπα, από τη στιγμή που λαμβάνει η χώρα καταστροφή μέχρι τις στιγμή όπου η περιοχή λαμβάνει τα κονδύλια. Από την άλλη, οι εθνικές περιφερειές και τοπικές αρχές οφείλουν ε, το ταχύτερο δυνατόν να επιταχύνουν και αυτά τις διαδικασίες τους. Κάτι άλλο θεωρώ ότι η κινητοποίηση του Ταμείου μπορεί να γίνει και μέσα από στενή συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, αυτούς δηλαδή που πλήττονται από την καταστροφή. Και κάτι άλλο. Θα ήθελα να παραθέσω αυτά τα οποία είπε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στη δική του γνωμοδότηση για το μέλλον του τραπείου, Ταμείου της Αλληλεγγύης. Αυτά έγιναν το 2012. Και όπως αναφέρει και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του του 15 Ιανουαρίου του 2013 σχετικά με την εφαρμογή του Ταμείου, Θέλω λοιπόν, παραθέτω η έκθεση αυτή, θέλουμε να καταδείξει ότι είναι απαραίτητο τα κονδύλια αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπληρώνονται και από άλλα κονδύλια όπως αυτά από τα διαρθρωτικά ταμεία. Να υπάρχει συνέργεια των διαφόρων μηχανισμών και αυτή η συνέργεια θα πρέπει όπως σας είπα να αφορά στα κονδύλια αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στα εθνικά ε, γιατί τα εθνικά κονδύλια, τουλάχιστον αυτά, δεν έχουν ακόμα δραστηριοποιηθεί. Άρα δηλαδή αυτό πλήττει την ανταγωνιστικότητα των περιοχών που έχουν πληγεί από την θεομηνία. Τελευταίο θέμα. Η πρόβλεψη παίζει καθοριστικό ρόλο ε, στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, θεωρούμε ότι μπορεί να βρεθεί ένας πιο οικονομικός τρόπος για να περιοριστεί το τροτό των περιοχών σε σχέση με τις θεομηνίες. Είναι απαραίτητο όλες οι περιοχές να χρησιμοποιούν με συνεπή τρόπο όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν έτσι ώστε να υπάρχει σωστή πρόληψη σε περίπτωση καταστροφών και μόνο αυτό αλλά και για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Αυτό που βιώνουμε τώρα αυτό είναι βασική αιτία που οδηγεί στις καταστροφές. Βεβαίω είμαι στη διάθεσή σα για να ακούσω τι δικέ σα προτάσει, ερωτήσει ε, και επιχειρήματα των συναδέλφων, των σκιωδών εισηγητών, αλλά και όλων των άλλων συναδέλφων τη Επιτροπής των Περιφερειών. Και δράτω με τι ευκαιρίε για να σα πω ότι ε, για του σκιώδει εισηγητέ, τις επόμενες εβδομάδε θα πρέπει να συναντηθούμε για να αξιολογήσουμε το κείμενο που θα μα έχει υποβληθεί. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τσίκου. Να ξεκινήσω με τους σκιώδες εισηγητές. Τον κύριο Πίκουλα. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όπως ακούσαμε, το Ταμείο Αλληλεγγύης συγκροτήθηκε για να παράσχει οικονομική στήριξη στα κράτη-μέλη και στις υποψήφιες χώρες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σε απάντηση στις πλημμύρες του 2002. και από την συγκρότησή του έχουμε ήδη καταβάλει 3,5 δις ευρώ μετά από 69 αιτήματα κρατών μελών και μη κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις αλλαγές που επιταχύνουν τη διαδικασία το 2014 και έτσι τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τέτοια κονδύλια σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Επίσης βελτιώθηκαν οι κανόνες για την επιλεξιμότητα των έργων. Και στόχος των ταμείων είναι να απαλύνουν τις, τον αρνητικό αντίκτυπο των φυσικών καταστροφών. Βασικό εμπόδιο είναι το ότι περνάει αρκετός ο χρόνος πριν να καταβληθούν τα κονδύλια, γιατί θα πρέπει να γίνει σωστή διοργάνωση και συνένεση μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου ενδεχομένως η χρηματοδότηση για τις πλημμύρες που ε, έπληξαν την Κροατία το 2014 το Μάιο δόθηκαν από την Κομισιόν τον Οκτώβριο και τις επικύρωσε το Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο μετά από 7 μήνες. Είναι κάτι που ε, πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά κατά τη γνώμη μου όταν μιλούμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Ένα άλλο θέμα είναι η αύξηση των κονδυλίων που φτάνουν τώρα μέχρι τα 100 εκατομμύρια. Θα πρέπει να αυξηθούν για να καλύψουν το εύρος της ζημιάς. Τα χρήματα που έχουν δοθεί έχουν καλύψει το 3-5% του συνολικού κόστους. Πρέπει να ενισχύσουμε την παρακολούθηση ε, αυτών των δαπανών. Σε κάθε περίπτωση περιμένω να συνεργαστώ με τους συναδέλφους για να έχουμε το καλύτερο δυνατό τελικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Πορέμπα είναι σκιώδης εισηγητής, αλλά δεν τον βλέπω στην αίθουσα. Ο κύριος Φαν Μίντελπορκ, που είναι επίσης σκιώδης εισηγητής για το Άλντε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Φυσικά Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τις φυσικές καταστροφές. Εξού και έχουμε το Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για να δείξουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με το πληγέν κράτος και την πληγή πληγήσα περιοχή. Σε κάθε περίπτωση η κάθε περιφέρεια ή το κάθε κράτος μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για να προλάβει τις καταστροφές και να περιορίσει ε, τα αποτελέσματά της. 8 δις για προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Η περιφερειακή πολιτική είναι στοιχείο κλειδί. Θα πρέπει οι περιφέρειες και τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για να προλάβουν τις φυσικές καταστροφές και να περιορίσουν τον αντίκτυπό τους. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, για κάθε ένα ευρώ που επενδύουμε για την πρόληψη, εξοικονομούμε από 4 έως 7 ευρώ στην ε, καταπολέμηση της βλάβης, της ζημίας. Επομένως, όλο αυτό είναι μια ευκαιρία για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης και μάλιστα βιώσιμες. Βεβαίως, σκοπός του Ταμείου είναι να, δώσει, να εκφράσει αλληλεγγύη και να βοηθήσει τους πληγέντες το συντομότερο, το γρηγορότερο δυνατό. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην έχει μεσολαβήσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι το ελάχιστο δυνατό το διάστημα από την έλευση της καταστροφής και την καταβολή της δαπάνης. Και θα πρέπει και τα κρατημέλη και το Κοινοβούλιο να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους έτσι ώστε να συντμηθεί η νομοπαρασκευαστική διαδικασία και έτσι ώστε να αξιοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι τα κονδύλια το συντομότερο δυνατό. Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές λόγω των μακροχρόνιων και μακροσκελών και διαπραγματεύσεων Συμβουλίου και Κοινοβουλίου πράγματα που έχουν συμβεί στην περίπτωση της Σαρδινίας π.χ. το 2013 είναι στοιχεία που υποδομεύουν την αποτελεσματικότητα του Ταμείου Αλληλεγγύης. Ωστόσο, άλλες χώρες και άλλες περιφέρειες που έχουν αξιοποιήσει τα κονδύλια του Ταμείου θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαίρως. Ε, και όλα αυτά θα βελτιώσουν τη διαφάνεια. Ελπίζω η αναθεώρηση που ξεκίνησε το 2014 με τον κανονισμό να επιταχύνει τελικά τη διαδικασία πληρωμών και να βελτιώσει την ορθή εφαρμογή και αξιοποίηση του περιεχομένου του Ταμείου Αλληλεγγύης. Ο αναθεωρημένος κανονισμός σίγουρα θα έχει αποτελέσματα, τα οποία όμως μπορούν να αξιολογηθούν μόνο τα επόμενα χρόνια και όχι σήμερα, γιατί θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα εμπειρίας. Ένα ένα σώμα ας πούμε, πυριών για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον να συνεργαστώ με τον εισηγητή. Η Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλους σκιώδεις εισηγητές εκτός από την κυρία Ντεμάτο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ε, μιλάμε για το Ταμείο Λεγγύης, για το κατά πόσο είναι απαραίτητο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω των θεμελιών και λόγω κλιματικών αλλαγών. Μιλάμε και για το Ταμείο αυτό που αφορά στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τις ε, μεγάλες καταστροφές, το Ταμείο Αλληλεγγύης μοιάζει να έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά, αλλά τα θέματα και τα ερωτήματα που αφορούν σε μικρότερες καταστροφές ε, ε, προκάλεσαν δυσκολίες σε κάποια κράτη-μέλη. Παραδείγματος χάρη, ο κανονισμός προβλέπει κάποιες προποθέσεις που είναι περίπλοκες. Ας πούμε, τα κράτη πρέπει να ορίζουν ακριβώς την περιοχή όπου επλήγησαν οι πολίτες, αλλά αυτό δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα. Γιατί για να αποδείξει κανείς ότι υπήρξαν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ε, στην οικονομική ζωή αυτής της περιοχής, αυτό είναι πολύ δύσκολο να το κάνει κανείς και για συγκεκριμένες περιοχές. Μέχρι τώρα ε, τα δύο τρίτα των ε, ετοιμάτων που κατατέθηκαν απορρίφθηκαν. Ε, είναι πολύ καλό που συζητάμε στην Επιτροπή αυτή αυτό το θέμα, το θέμα της, ε, του Ταμείου Αλληλεγγύης, αλλά πρέπει να το κάνουμε κάτω από το πρίσμα ότι πρέπει να περιοριστούν οι δυσκολίες, αλλά και η βραδύτητα που επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση των ετοιμάτων πρέπει να συνεργαστούμε στενά για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Και από την άλλη πρέπει να πούμε ότι αν τελικά τα κονδύλια αυτού του ταμείου ε, δεν δόθησαν ε, σε περιπτώσεις που θα έπρεπε, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να βελτιώσουμε το καλό και να αποκλείσουμε τις ε, καταχρήσεις και τις περιπτώσεις εγκληματικών ενεργειών. Θα ήθελα να φέρω ως παράδειγμα, ε, οι εκθέσεις που, κατατίθενται από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτές. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υλοποιηθούν μέτρα έστω προσωρινά σε περι... Περιοχέ που έχουν καταστραφεί. Και θα ήθελα να φέρω ένα παράδειγμα το οποίο αφορά τη δική μου τη χώρα και να σα υπενθυμίσω ότι δεν δόθηκε καμία συνέχεια στι ανησυχίε που εκφράστηκαν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την χρήση των κοντιλίων στην περιοχή Αμπρούτσο. Ε, Εκεί υπήρχε ένα σχέδιο για την κατασκευή κατοικιών ε, και δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα, ε, ελληματικά ε, υλικά και κάποια μπαλκόνια μάλιστα κατέρευσαν, αυτό το είδαν όλοι. Ως εκ τούτου, για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά, θέλουμε να συνεργαστούμε με τον εισηγητή και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα λάβει και αυτό στις δικές μας απόψεις, στη δική του την εισήγηση. Η πρόεδρος εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα ήθελα να υποφεληθώ για να πω με δύο λόγια την άποψή μου και να κάνω και μια πρόταση. Θα ήθελα στην έκθεση του κυρίου Τσίκου να σταθμίσουμε το μέγεθος των ζημιών και το χρόνο καθυστέρησης. ενάμιση χρόνος ήταν στη Σαρδινία για παράδειγμα. Αυτή η καθυστέρηση θα πρέπει σίγουρα να συνημηθεί και να κάνουμε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Είδαμε τι έγινε στο Εμιλιό. Για μερικές... Είναι... Ε, ξέραμε ότι η καταστροφή είχε γίνει και παρόλα αυτά η Κομισιόν δεν πρέπει να πληρώμες. Θα έπρεπε να έχει ε, τη διακριτική ευχέρεια η Κομισιόν να μπορεί να κάνει προκαταβολές, ε, σημαντικές ε, προκαταβολές, ο, μόλις γίνει η καταστροφή, γιατί αν να περιμένουμε ένα, ένα μισή χρόνο είναι πια πολύ καθυστερημένο. Είδα στην Κροατία για παράδειγμα, το παράδειγμα, ε, στην Κροατία έφτασε είναι πολύ μικρό ποσό αμέσως, πολύ μικρό, ελάχιστο, σήμαντο. Θα πρέπει αυτοί που έχουν πληγεί, πληγέντες, να μπορούν να εισπράττουν κάποια ποσά, όχι τεράστια ποσά, ένα αξιοπρεπές ποσό όμως, αμέσως. Γιατί η μία πρώτη αξιολόγηση μπορεί να γίνει στις πρώτες δέκα μέρες. Και μπορούμε πλέον να ξέρουμε αν οι ζημιές ήταν σημαντικές ή όχι και να πληρώσουν τα αντίστοιχα ποσά 10-15% των ζημιών. Αλλιώς περνάει χρόνος πολύ και ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι κανείς δεν, λαμβάνει, δεν τους λαμβάνει υπόψη. Αντιθέτως, αν οι πληρωμέ γίνουν αμέσω φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει αλληλεγγύη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, κ. Μάνσκο. Ευχαριστώ τον εισηγητή να υπογραμμίσω το πόσο το Ταμείο Συνοχής είναι απαραίτητο. Είναι ένα από τα πιο γλαφυρά παραδείγματα των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται. 600 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται σε αυτό το ταμείο κάθε χρόνο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή. Το ταμείο αυτό έχει ως προτεραιότητα βέβαια τις θεομηνίες σε εθνικό επίπεδο ε, αλλά χαίρομαι που είναι δυνατόν να κινητοποιηθεί και σε περιφερειακό επίπεδο. Χάρη στην ε, εργασία που έγιναν στην περασμένη κοινοβουλευτική θητεία. Εγώ προέρχομαι από υπερπόντιο διαμέρισμα και χαίρομαι που η, ε, που καλύπτονται επαρκώς οι ε, άκρως περιφερειακές, περιφερειακές, ε, εξόχους τη περιοχές της κοινότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι ε, ε πλήττονται πολύ συχνά από θεομηνίες και ε, που όμως δεν είναι εθνικού μεγέθους, εθνικού βεληνικούς, δεν αναγνωζόντουσαν στο παρελθόν ως δικαιούχες περιοχές. Τώρα πια μπορεί το Ταμείο να κινητοποιηθεί αν οι καταστροφές ε, καλύπτουν ε, το 1% του ΑΕΠ της συγκεκριμένης ε, περιοχής. Ε, χαίρομαι για, αυτό, για αυτή την αλλαγή. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν το λόγο. Ο κ. Τσίκου. Πριν από εσάς όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρω αν ε, αντιπροσωπεύεται. Θέλει το λόγο. Ορίστε. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο. Ε, έχουμε απεργία στα μέσα συγκοινωνίας και έχει πολύ κίνηση στο δρόμο. Οπότε δεν άκουσα τον, την αρχική εισήγηση του εισηγητή, λυπάμαι πολύ. Πριν όμως να υπογραμμίσω ότι η Κομισιόν ενδιαφέρεται πάρα πολύ, είναι πολύ πρόθυμη να συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή σας και με τον εισηγητή. Σε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας. Και νομίζω ότι μπορούμε να προσφέρουμε διευκρινήσεις και λεπτομέρειες που θα είναι χρήσιμες για την έκθεση να επαναλάβω κάτι που υπόθηκε και προηγουμένως. Ε, πράγματι αναθεωρήθηκε ο κανονισμός για το Ταμείο Συνοχής της Ελληνικής, συγγνώμη, πριν από δύο χρόνια. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι λίγο πρόωρο να βγάλουμε συμπεράσματα, να κάνουμε μια αξιολόγηση. Η τελευταία περίοδος, η τελευταία διετία δεν χαρακτηρίστηκε από πάρα πολλές θεομηνίες. Ε, από το 2014 και μετά, 12 συνολικά, εκ των οποίων οι περισσότερε ε, έλαβαν χώρα στο τέλο του 2014 και 2 μέσα στο 2015, συγγνώμη το 2016. Οπότε στατιστικά δεν είναι πολύ μεγάλο το δείγμα για να βγάλουμε συμπεράσματα. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμω είναι ότι τα νέα κριτήρια για τι ε, τοπικές ε, θεομηνίες ε, σε επίπεδο περιφέρεια δηλαδή είναι πλέον πολύ πιο σαφή. Βέβαια, προ το παρόν δεν έχουμε ε, αιτήματα για τέτοιου είδου θεομηνίες ακόμα. Μάλλον δεν έχουμε απορρίψει κανένα τέτοιου είδου αίτημα και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον αυτή η τάση ε, ελπίζουμε ότι η, ο δείκτης αποδοχής των ετοιμάτων θα είναι περίπου 100% όπως και μέχρι τώρα ε, έτσι ώστε να καλύπτουν πραγματικά όλες τις μείζων σημασίας καταστροφές ε, όπως είναι και ο στόχος του Ταμείου. Συνολικά είναι λογικό να πούμε ότι το Ταμείο έχει λειτουργήσει αρκετά ικανοποιητικά 102 αιτήματα έχουν ληφθεί από το 2002 70 εγκρίθηκαν όλες οι απορρίψεις αφορούσε σχετικά μικρές τοπικές θεομηνίες που ελπίζουμε ότι στο μέλλον δεν θα απορρίπτονται και τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν ε, ήταν το συνολικό κονδύλι ε, του Ταμείου που έχει δαπανηθεί ως τώρα. Ε, τώρα για ορισμένα θέματα που εθίξαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Αυτή τη στιγμή πλέον έχουμε πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια, ευκρίνεια σε ό,τι αφορά τις ε, θεομηνίες, τις ε, ε, ε περιοχές. Ε, έχουμε ένα κατόφλι χαμηλότερο από τις υπόλοιπες περιοχές, περιφέρειες. Αυτό εξαιτία του γεγονότου του χαρακτήρα των περιοχών αυτών που εκτίθενται περισσότερο στις ε, θεομηνίες, είναι πιο εκτεθειμένες. Η Κομισιόν συμφωνεί απόλυτα ότι θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να συντμίσουμε το χρόνο ε, ανάμεσα στην θεομηνία και την πληρωμή των ενισχύσεων. Όπως γνωρίζετε, ο καινούριος κανονισμός ε, προβλέπει μια διαβριμένη περίοδο ε, αίτησης αιτήματος, τις 10 περνάμε στις 12 εβδομάδες και γενικά τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν πλήρω αυτή την ε, περίοδο, οπότε υπάρχει ήδη μια πρόσθετη καθυστέρηση δύο εβδομάδων. Απ' την άλλη μεριά, οι διηγητικέ διαδικασίε έχουν συνδυμηθεί σε κάποιο βαθμό, οπότε αν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ω Δημοσιονομική Αρχή δεχτούν όποτε ε, δέχονται του ε, συμπραγματικού προπολογισμού προκειμένου να κινητοποιηθεί το Ταμείο το Συντομότερο Δυνατό, αυτό, από αυτό εξαρτάται ε, και η ταχύτητα. Επίσης προβλέπει ο κανονισμός ε, τη δυνατότητα να δίδονται προκαταβολές, ε, θίγει αυτό που κάποιον από τους ομιλητές, 10% συνολικά του αναμενόμενου ποσού ενίσχυσης. Το αναμενόμενο ποσό ενίσχυσης βέβαια δεν καλύπτει όλες τις ζημιές μιας θεομηνίας, όπως γνωρίζετε, με 500 εκατομμύρια που έχουμε κάθε χρόνο διαθέσιμα δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε με πολύ ψηλά ποσά. Βέβαια, για του Δήμου τι κοινότητες, για τι περιφέρειες και τα κρατημέλη είναι σημαντικά ποσά, αλλά σίγουρα δεν αποζημιώνουμε το σύνολο των ζημιών. Έχουμε χρησιμοποιήσει αυτή την ρυθμίση, αυτή την μέρημνα του νόμου από την, ε, από την αρχή του 2015 στις τρεις από τις τέσσερις περιπτώσεις για τις οποίες έχουν γίνει έκτοτε έχουν κατατεθεί αιτήματα ε, η πρόβλεψη αυτή χρησιμοποιείται μόνο όταν μας ζητηθεί. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε την χρήση της, ε, μάλλον θα, για τον Ηνωμένο Βασίλειο στην τελευταία του αίτηση δεν ζήτησε να χρησιμοποιηθεί αυτή η διευκόλυνση της προκαταβολής, γι' αυτό το λόγο και δεν θα χρησιμοποιηθεί. Ε, αυτά είχα να πω για την έκθεση. Δεν ξέρω αν έχετε άλλες ε, ερωτήσεις. Είμαστε στη διάθεσή σας. Thank you, thank you very much. And now... Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίκου. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές ότι κατέγραψα όλα αυτά που ελέγχθησαν από τους συναδέλφους. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την άποψη της Επιτροπής και θα έχουμε και τη συνάντηση με τους σκιώδης ηγητές έτσι ώστε να έχουμε μία σφαιρική άποψη στην οποία θα καταλήξουμε. Ευτυχώς η περιπτώσεις ε, που ήταν πολύ κρίσιμες ήταν πάρα πολύ λίγες. Αυτό σας λέω ευτυχώς. Παρ' όλα αυτά πρέπει να αξιολογήσουμε τις περιπτώσεις αυτές και νομίζω ότι ε, όταν θα το κάνουμε αυτό θα είναι μια πολύ καλή συνεισφορά αυτής της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ήταν η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Εξ όσων γνωρίζω, ο κύριος Τσίκου θα παρουσιάσει το προσχέδιο έκθεσης του στη συνεδρίασή μας τον Ιούλιο και θα το ψηφίσουμε το Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε την εξέταση αυτού του σημείου της ημερήσιας διάταξης. Επόμενο σημείο είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Γιουίρκη Κατάινεν, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, επιφορτισμένος με το χαρτοφυλάκιο ε, για την απασχόληση, την ανάπτυξη, την επένδυση και την ανταγωνιστικότητα. Δεν έχει έρθει ακόμα θα πρέπει να περιμένουμε 15 λεπτά. Έχετε 15 λεπτά να τα αξιοποιήσετε όπως θέλετε. Είναι όντως ώρα για έναν καφέ. Ladies and gentlemen, can I ask for your attention, Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ την προσοχή σας. Ακριβώς στις 4.30 ξεκινούμε. Ο κύριος Κατάινεν, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βρίσκεται στην αίθουσα και μετέχει στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Με χαρά τον καλωσορίζουμε έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των υποθέσεων για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βρίσκεται στην Επιτροπή μας για να συζητήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών επενδύσεων και τις συνέργειες που έχει με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, αλλά και τις λοιπές πτυχές της πολιτικής συνοχής που συνδέονται με το δικό του χαρτοφυλάκιο. Τον Μάρτιο του 2015 τον συναντήσαμε την περασμένη φορά. Εκείνη την ε, ημέρα είχε πάρει το λόγο μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής αλλά και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να μας παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ΕΦΣΥ. Και η σημερινή του παρουσία εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής εξέτασης της Ευρωπαϊκής Διαδικασίας. Ήταν Υπουργό Οικονομικών και ε, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Φιλανδίας. Θα δώσω το λόγο στον αντιπρόεδρο και θα ξεκινήσει η συζήτηση. Στη συνέχεια θα πάρουν το λόγο οι συγητές. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε για ό,τι θέλετε. Μπορώ Ίσως να προσπαθήσω να δώσω απάντηση σε όλα σας τα ερωτήματα. Ε, σήμερα αυτό που μας απασχολεί είναι η υλοποίηση του προγράμματος εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουμε βέβαια πολλούς, ε, πολλές ε, επικεφαλίδες και υποτίτλους σε κάθε κεφάλαιο. Όμω, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τι επενδύσεις κυριαρχούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ΕΦΣΥ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων τα πηγαίνει πολύ καλά. Τα project, τα έργα για την εσωτερική αγορά επίσης πηγαίνουν καλά. και θα αποκαλύψουμε και το, την ευρωπαϊκή πύλη, το πόρταλ για τα ευρωπαϊκά έργα και μπορούμε και να ε, συζητήσουμε περισσότερο γι' αυτό αν σας ενδιαφέρει, γιατί θα είναι λειτουργικό από 1η Ιουνίου. Επίσης, τα συμβουλευτικά έργα για τις περιφέρειες και τα κράτη ε, λειτουργούν και προχωρούν. Έχουμε διάφορα θέματα που συνδέονται με την ενιαία αγορά. Η Συμφωνία για το Κλίμα των Παρισίων, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η κυκλική οικονομία, η περαιτέρω ανάπτυξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εκτός των άλλων. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω με την πολιτική συνοχής. Με προπολογισμό 450 δις ευρώ από το 2014 μέχρι το 2020, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων αποτελεί και το βασικό εργαλείο επενδυτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βελτιώσει και να ενισχύσει τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων με ε, ενδιαφέρον και έμφαση στα αποτελέσματα θέλουμε να έχουμε επενδύσεις σε παιδεία που βασίζονται σε καλό στρατηγικό ε, σχεδιασμό και να συνδέσουμε τις επενδύσεις σε ε, διάφορα προαπαιτούμενα που συνάδουν με τη στρατηγική μας. Όλα αυτά συνάδουν και με το ευρωπαϊκό ε, εξάμεινο, με τις, ειδικές, με τις ειδικές συστάσεις αναχώρα μεταξύ άλλων. Η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων εξαρτάται από υγιείς δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να ενισχύσει την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για να στηρίξει τις βασικές προτεραιότητες που τονίζονται στις ειδικές συστάσεις αναχώρα συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση. Τα κονδύλια αυτά δεν θα ανασταλούν λόγω της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος παρά μόνο σε, ε, στην περίπτωση απουσίας δράσης από πλευράς κυβερνήσεων για να επιληθούν αυτά τα θέματα. Ο συνδυασμός ΕΦΣΙ και ΕΣΥΦ είναι εφικτός και μπορεί να γίνει και σε επίπεδο έργου, αλλά και σε επίπεδο επενδυτικής πλατφόρμας, εθνικής, κλαδικής ή περιφερειακής. Και πρέπει να συνεργαστούμε ακόμη πιο στενά για τα ζητήματα αυτά. Οι περιφέρειες δεν γνωρίζουν αυτές τις ευκαιρίες ακόμα. Εσείς εκπροσωπείτε τις κοινότητες, τους λαούς, τις περιφερειές και διαδραματίζετε πολύ σημαντικό ε, ρόλο. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε, έτσι ώστε οι περιφερειές σας να βρουν ευκαιρίες να συνδυάσουν κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων με κονδύλια από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για να υλοποιήσουν έργα που ε, θα τις βοηθήσουν. Ο συνδυασμό στήριξη από τα διαφορετικά αυτά ταμεία κομίζει προστιθέμενη αξία και για τα δύο. Με το ΕΦΣΥ έχουμε αυξημένο όγκο κονδυλίων, ενώ το ΕΣΥΦ επιτρέπει στο ΕΦΣΥ να αναλάβει υψηλότερο κίνδυνο και άρα να προσελκύσει ακόμα μεγαλύτερους επενδυτές. Έχουμε δημοσιεύσει ένα φυλάδιο για την αλληλοσυμπληρωματικότητα μεταξύ αυτών των δύο εργαλείων για να ενημερώσουμε τα εμπλεκόμενα μέρη για τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που έχουν. Και σύντομα θα έχουμε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα του πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα στην πράξη. Το πρώτο έργο που υλοποιείται είναι στη Βόρεια Γαλλία, εάν δεν με απατά η μνήμη μου. Και είναι εύκολο να αναδειχθεί ως παράδειγμα και για τους υπόλοιπους. Η προγραμματική περίοδος 2014-2020 θέλει να αξιοποιούμε ε, χρηματοπιστωτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία για να ενισχύσουμε τις επενδύσεις. Αυτό είναι βασικό στοιχείο του ΕΦΣΥ. Τονίζεται η ανάγκη μεγαλύτερο μερίδιο του ΕΣΥΦ να δαπανάται μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών και χρηματοπιστωτικών ε, εργαλείων. Έχουν διπλασιαστεί, ε, στόχος είναι να διπλασιαστούν αυτά από το 2014 μέχρι το 2020. Είναι, αισιόδοξο αλλά ρεαλιστικό. Άνω των 20 δις ευρώ είναι ο φάκελος ο χρηματοδοτικός διπλάσιο σχεδόν από το 11,5 δις ευρώ της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας δώσω το παράδειγμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο ΕΤΠΑ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης δίδεται η στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η Επιτροπή ενθαρρύνει να μεταφέρουμε αυτή τη στήριξη στα χρηματοδοτικά και χρηματοπιστωτικά εργαλεία για διάφορους λόγους. Η, ε, γίνεται μόχλευση περισσότερων πόρων, άρα ο αντίκτυπος είναι πολύ σημαντικός. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το βασικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις άμεσες ενισχύσεις είναι ότι δίδεται ενίσχυση πριν γίνει η επένδυση. Αξίζει να αναφερθεί και η πρωτοβουλία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διοχετεύει το ΕΣΥΦ στο ΕΦΣΥ. Έχει σχεδιαστεί ως ένας μηχανισμός αποτελεσματικότητας για να έχουμε επιπρόσθετο δανεισμό από τον τραπεζικό τομέα η Ισπανία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ιταλία αλλά και η Φιλανδία έχουν συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι σήμερα. Ε, δύο λόγια να σας πω για την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Καταρχάς, να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τη διαδραμάτιση ρόλο κλειδί κατά τις διαπραγματεύσεις ε, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και προέβλεψε για επαρκή ευελιξία, η οποία ε, λειτουργήσε ως εργαλείο το 2014 για να στεθεροποιήσουμε το backlog, το, το τέλμα των καθυστερούμενων πληρωμών της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου. Και συμφωνήσαμε σε κοινή δήλωση για ένα σχέδιο πληρωμών έτσι ώστε μέχρι το 2016 να μειωθεί το ύψος των απλήρωτων λογαριασμών σε ένα βιώσιμο επίπεδο. Η ενδιάμεση αξιολόγηση, η ενδιάμεση ε, αναθεώρηση θα μας δώσει την ευκαιρία να εξετάσουμε αυτές τις λειτουργίες και να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον προϋπολογισμό πιο αποτελεσματικά για να ανταποκριθούμε στις βασικές κρίσεις. Δεν αποφασίσαμε ακόμα για τις προτάσεις μας για τον τίτλο των προτάσεων μας για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Αυτό θα το κάνουμε ε, στο εύρος αυτής της, ε, κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς. Ωστόσο, διάφορες προσδοκίες αντιβαίνουν, αντι, παρέρχονται μία την άλλη. Άλλοι θεωρούν ότι θα υπάρξουν, αύξηση, ε, θα υπάρξουν αυξήσεις στις επενδύσεις. Άλλοι δεν επιθυμούν να στηρίξουν την αναθεώρηση. Κάθε αναθεώρηση απαιτεί από το Συμβούλιο να αποφασίσει ομοφόνος, έχοντας αποκτήσει την συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι ευρεία είναι η συνένεση για την ποιοτική διάσταση του θέματος. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή περισσότερη ευελιξία και περισσότερη απλούστευση κατά την εφαρμογή όλων αυτών. Ήδη έχουμε εξαντλήσει το περιθώριο ευελιξίας μας, το υφιστάμενο, για να αντιμετωπίσουμε διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η προσφυγική κρίση. Η νομοθετική ε, πρόταση για την απλούστευση των εργαλείων ευελιξίας θα αποτελέσει μέρο της δέσμη των προτάσεων αυτών. Έγινε διαβούλευση με ε, διάφορους φορείς στις αρχές του Μαρτίου για να συμμορφωθούμε με τους κανόνες για καλύτερη νομοθέτηση. Και άλλωστε γίνεται και δουλειά ε, σε, με αυτή την πρωτοβουλία σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός πρέπει να δίνει έμφαση στα αποτελέσματα. Με αυτά τα δύο κριτήρια έγινε η συζήτηση με το Συμβούλιο. Και θα πρέπει να αναθεωρηθούν για το 2017 οι σχετικοί φάκελοι για τις περιφέρειες που αφορούν στις περιφέρειες μέσα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Μιλούμε ε, για τις οροφές, τα κατόφλια ε, πληρωμών και δαπανών και πιστώσεων που ε, αποφασίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τεχνικό δελτίο. Πολλά από αυτά θα πρέπει να έχουν λυθεί με το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα καθορίσουν και την πρόταση που θα διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, την οποία και θα παρουσιάσει τον Ιανουάριο του 2018. Ως προς τους ίδιους πόρους και το μέλλον αυτών, περιμένουμε να ολοκληρώσει τις συστάσεις της η ομάδα υψηλού επίπεδου για το θέμα αυτό υπό την προεδρία του κυρίου Μόντι. Και το σημαντικό θα είναι η διακοινοβουλευτική ε, διάσκεψη που προγραμματίζεται για το Σεπτέμβριο του 2016 φέτος. Παρακολουθούμε το έργο της ομάδας υψηλού επίπεδου επίσης για την απλούστευση. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου να ενσωματώσουμε κάποια από τα συμπεράσματα της ομάδας αυτής. Να σας εφιστήσω την προσοχή σε αυτό το θέμα, το οποίο ε, ανταποκρίνεται σε πολλές διεκδικήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρίως το έχετε θέσει αυτό το θέμα στην Επίτροπο Κρέτσου. Και θα ήθελα να, προσθέσω ότι ε, το προγραμματικό πλαίσιο, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, έτσι όπως εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή, η εφαρμογή του είναι που ε, μας κάνει να θέτουμε τα ζητήματα που χρήζουν βελτιώσεων. πρέπει το 5% ε, των ετοιμάτων πληρωμής ε, έχει κατατεθεί φέτος για το σύνολο της χρονιάς σε σχέση με αυτό που είχε προβλεφθεί. Πρέπει να έχουμε σωστή εφαρμογή, σχεδιασμό και προγραμματισμό. Πρέπει να η προπαρασκευαστική εργασία επαρκής. Και μετά από αυτά Ήδη το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τα κατάλληλα κείμενα, παρόλο που είχαν σημειωθεί καθυστερήσεις στο παρελθόν. Το πλαίσιο λοιπόν δίνει έμφαση στα αποτελέσματα και η εραρχή της επενδύσης, έτσι ώστε να χρηματοδούν επαρκώς τα προηγούμενα έργα που είχαν ήδη εγκριθεί. Όμως, η εφαρμογή των έργων, τα προγράμματα εφαρμόζονται υπό την ευθύνη των κρατών μελών. Έχουμε μοιρασμένη τη διοίκηση, τη διαχείριση όλων αυτών των έργων και γι' αυτό είναι πιο αργή η ρυθμή, ειδικότερα ως προς τις ενδιάμεσες πληρωμές, την ικανοποίηση όλων αυτών των σχετικών ετοιμάτων. Υπάρχει καθυστέρηση στον ορισμό των διαχειριστικών αρχών έργου από τα κράτη-μέλη και αυτό είναι προαπαιτούμενο προϋπόθεση για να εγκριθούν οι ενδιάμεσες προσωρινές αιτήσει πληρωμής δαπανών. Και όλα αυτά βεβαίως μπορεί να συνθέονται με τα προαπαιτούμενα, την αιρεσιμότητα εξάντε και ενίοτε ε, κάθε φορά που έχουμε ελέγξει τις προϋποθέσεις μπορεί να έχουν συμβεί περιπτώσεις όπου έχουμε αποφασίσει την αναστολή γιατί υπήρχαν προβλήματα εκεί. Τέλος, θα ήθελα να πω και δύο λόγια για την προσφυγική κρίση, η οποία έχει αλλάξει τις προτεραιότητες στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. δεν έχει υποβληθεί κάποια τροποποίηση για κάποιο εθνικό ή περιφερειακό έργο. Καλεί η περιφερειακο εργο Καλή επιτροπη ομως τα κράτη-μέλη να επανεξετάσουν τον προγραμματισμό τους από το 2014 μέχρι το 2020 για να δουν κατά πόσο ε, μπορούν να ενισχυθούν κάποια μέτρα που να έχουν να κάνουν και με την προσφυγική κρίση. Το ΕΤΠΑ μπορεί να χρηματοδοτήσει πολλά και διαφορετικά, πολλές και διαφορετικές δράσεις, στέγαση, υποδοχή, ε, δίκτυα ίδρευσης, ε, εκπαίδευση, υγεία, μεταξύ άλλων. Η μετανάστευση είναι μια πραγματικότητα στα αστικά κέντρα, και θα πρέπει οι πόλεις να αντλούν τα διδάγματα η μία από την εμπειρία της άλλης, εντάσσοντάς τα στην ευρωπαϊκή προοπτική. Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για Καινοτόμες Δράσεις ζητά να υποβλεθούν προτάσεις για την καλύτερη διαχείριση ε, των ροών μεταναστών και προσφύγων για την καλύτερη συνέργεια όλων των οργανώσεων, δημόσιων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, Επομένως, οι, οι, εκδηλώσεις στο Άμστερνταμ θα είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα αστικά κέντρα. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Πρόεδρε, είμαι στη διάθεσή σας και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα για ε, τα θέματα διαρθρωτικής πολιτικής και επενδύσεων. Είναι μια ευκαιρία να μάθω και από εσά, να ακούσω τις εμπειρίες σας Και αν σας ενδιαφέρει, μπορώ να σας ε, αναπτύξω ε, τις ευκαιρίες που υπάρχουν με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Τι έχουν κάνει οι άλλοι και τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Ευχαριστούμε. Κύριε Αντιπρόεδρε, είμαι σίγουρο θα ακούσετε πολλά για την πολιτική συνοχή, για τη μελλοντική πολιτική συνοχή, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, για το μελλοντικό πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Όλα αυτά τα θέματα είναι στην, στα, μεταξύ των ενδιαφερόντων μα και είμαι σίγουρος, ότι θα τεθούν πολλά ερωτήματα. Ξεκινάμε με ερωτήσεις λοιπόν και προτάσεις από τους συντονιστές. Καταρχήν ο κ. Φαν Νίστελροϊκ, εκ του ΕΛΚ. Καταρχήν θέλω να σας συγχαρώ. Γιατί είστε ε, ε, έξοχος στην ε, χρήση των μέσων επικοινωνίας. Βλέπω τα tweets σας, βλέπω ε, τις ανακοινώσεις, ε, τα ανακοινωθέντα τύπου. Βλέπω τις καθημερινές ενημερώσεις στο site σας κλπ Τώρα είπατε ότι το, το πρώτο αυτό πράγμα που θα μπορούσαμε να κρίνουμε θα φτάσει ίσως τον Ιούνιο. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, δεν κατάλαβα πολύ καλά. Ε, εμείς στον κανονισμό για το ΕΦΣΥ είχαμε πει ότι είχαμε συμφωνήσει ε, να εξετάσουμε τι συνέργειες θα δημιουργηθούν. Ήταν καινούριο, δεν ξέραμε ποιο θα ήταν το μέλλον του ακριβώς. Ήταν δύσκολο να προβλέψουμε ε, την διείσδυσή του. Και είχαμε πει ότι μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσουμε τον κανονισμό αν χρειαστεί. Οπότε και εμείς είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι όπως και εσείς, αλλά περιμένουμε περισσότερα αποτελέσματα. Εγώ διαφημίζω το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, παντού όπου σταθώ και όπου βρεθώ. Και αν χρειαστεί θα κάνουμε και νομικές αλλαγές τροποποίηση στον κανονισμό του. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, σε, ό,τι αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το ΕΛΚ, ε, λέει ότι ε, δισεκατομμύρια ε, ευρώ που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ε, να μην επιστρέφουν στα κράτη-μέλη. τώρα αυτό συνέβαινε. Ε, όλο, συνεχώς ζητούμε φρέσκα χρήματα ε, για την γεωργία παλιότερα, για την περιφερειακή πολιτική, ε, ενώ στην πραγματικότητα τα έχουμε. Αντί να ζητάμε λοιπόν από τα κράτη-μέλη, ας μην τους επιστρέφουμε το υπόλοιπο. Το μη αναλωθέν υπόλοιπο του προπολογισμού. Αυτό είχαμε πει μαζί με τον κύριο Όλμπριχτ που ήταν συνσύγητης. Αν μιλάμε για ευελιξία, ανάμια ευελιξία είναι κοινωτικά χρήματα. Και για τους πρόσφυγες μπορούμε να κάνουμε πολλά. Είναι, αυτά είναι χρήματα που έχουμε και αρμοδιότητα την οποία διαθέτουμε. Δεύτερο ήταν αυτό. Τρίτο. Είστε πρωταθλητής στην πολλαπλασιαστικότητα. Εμείς λέμε ότι κάθε ευρωπαϊκό ευρώ πολλαπλασιάζεται επί τέσσερα τελικά. Εσείς τι είχατε πει, 20? Ε, και περισσότερο λέτε ο πολλαπλασιαστής σας είναι ακόμα μεγαλύτερος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον. Εμείς έχουμε πλέον μια μελέτη που δείχνει πού χρειάζεται η δωρεάν βοήθεια, ε, η επιδότηση. Οι κρατικές δομές, η έρευνα, εκεί που κανείς άλλος δεν θέλει να επενδύσει. Ε, γιατί στους άλλους τομείς ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, εργαλεία της αγοράς και να προσετεριστούμε επενδυτές. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μας λέει αυτά που μας έλεγε πάντοτε, αλλά δεν αρκεί. Δεν αρκεί αυτό. Αν τα 20 γίνουν 40, πού θα τελειώσουμε στην επόμενη περίοδο. Θέλω να συζητήσουμε σοβαρά με το Συμβούλιο, με όλους τους εμπειρογνώμονες για αυτό το θέμα. Και τέλος, ποια είναι η σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη. Μόλις γύρισα από την Σλοβενία και την Κροατία. Τον Περνό μήνα μάλλον πήγα εκεί. Και Τα νέα κρατημέλη, στα οποία επενδύουμε πολλά κονδύλια της περιφερειακής πολιτικής, εξακολουθούν να υστερούν. Πολύ. Και δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα από αυτά που γίνονται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν έχουν την κατάλληλη ορμή, την ταχύτητα που χρειάζεται για να εκμεταλλευτούν όλες τις δυνατότητες που δίδονται. Δεν έχουν τις ικανότητες και μετά την κρίση βλέπω ακόμα μεγαλύτερες διαφορές. Και αυτό δεν είναι θέμα πρόβλημα της συνοχής του α ή του β. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Οπότε το ερώτημα είναι τι θα γίνει μετά από αυτήν την περίοδο. Οι περιφέρειες σύγκλησης έλαβαν μια σημαντική όθηση Εκεί έχουμε τρεις σταυρούς, τρία συν, ένα ακόμα στα παλιά κράτη-μέλη, 65% του ορίζοντο 2020 είναι στα παλιά κράτη-μέλη και πολύ λιγότερο στα νέα κράτη-μέλη. Τι γίνεται τώρα εκεί. Ελπίζω ότι με τον ΕΦΣΥ ε, θα βελτιωθεί η κατάσταση και ότι θα το συζητήσουμε τουλάχιστον. Χρειαζόμαστε περισσότερη ελεγγύη. και ελπίζω ότι η πρότασή σας θα είναι ισορροπημένη. Εσείς λέτε είμαστε εντάξει αυτή τη στιγμή σε σχέση με τους στόχους μας. Ευχαριστώ κυρία Κρέιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχω κάποια ερωτήματα που αφορούν στην πολιτική συνοχή και κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα. Όσον αφορά την πολιτική συνοχή, εγώ ισχυρίζομαι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαπραγματευτεί μια πολύ καλή πολιτική συνοχή η οποία ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις. Εσείς τι πιστεύετε, συμφωνείτε μαζί μου. Ε, και το ρωτάω αυτό με απόλυτη ακρίβεια, γιατί ξέρετε, ακούω ε, επανειλημμένα ε, φήμες από την Κομισιόν, όχι απαραίτητα από τη δική σας τη Γενική Διεύθυνση, που λένε οι φήμες αυτές ότι η πολιτική συνοχή είναι πλέον παντελώς παροχημένη, δεν τη χρειαζόμαστε καν. Καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα του Juncker με μόχλευση 1 προς 17 και θα τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα. Το δικό μου λοιπόν το ερώτημα είναι, εσείς με τι συμφωνείτε, με αυτή την άποψη ή με την άποψη ότι χρειαζόμαστε μια σύγχρονη ε, πολιτική συνοχή για το μέλλον. Το δεύτερο ερώτημά μου είναι το εξή. Υπάρχουν άραγε προγράμματα όπου να διαφαίνεται ότι πράγματι προκύπτει αποτέλεσμα από τη μόχλευση όπως είχε προβλεφτεί. Θα χαιρόμουν να συμφωνήσετε, αλλά έχω κάποιες αμφιβολίες. Τρίτο ερώτημα. Το τίξατε κι εσείς. Μιλήσατε για την μακροοικονομική αιρεσιμότητα, όπως αποκαλείται. Το Κοινοβούλιο ήταν ανέκαθεν κατά αυτού, τουλάχιστον η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τελικά το δεχτήκαμε πράγματι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Πρέπει κανείς να κάνει συμβασμού και τώρα υπάρχει αυτή η μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Εσείς τι πιστεύετε, υπάρχουν εξελίξεις που να αποδεικνύουν ότι είναι καλό που υπάρχει αυτή η αιρεσιμότητα, ε, γιατί έχει άμεση σχέση με τις μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Και με ενδιαφέρει το κατά πόσο να έχετε πληροφορίες επ' αυτού. Επίσης, και κάτι άλλο, πιστεύω ότι οποτεδήποτε στηρίζουμε τα χρηματοοικονομικά μέσα για την πολιτική συνοχής. θα πρέπει να αποδεικνύουμε γιατί το κάνουμε αυτό. Θα πρέπει αυτά ίσως να παραμένει βάση της πολιτικής μας, γιατί ξέρετε, ε, δεν μπορώ να πω ότι αυτά τα μέσα και γενικότερα η πολιτική θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο με δανειοδοτήσεις, αφού και πρέπει να υπάρχουν και επιδοτήσεις. Είναι ένα θέμα επίμαχο. Όσον αφορά την ενδιάμεση αναθεώρηση του, ε, του ε, μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου έχουμε καταρτήσει μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή μας και ένα πράγμα είναι απόλυτα σαφές ότι δεν επιθυμούμε να υπάρξει περικοπή των ε, κονδυλίων συνοχής. Γιατί αυτά είναι χρήματα των φορολογουμένων που έχουν επενδυθεί πολύ σωστά. Αλλά ξέρετε, πολλοί λένε, μα έχουμε τόσα πολλά χρήματα που μπορούμε να δώσουμε και κάτι, να λύσουμε και το α και το β και το γ πρόγραμμα ή πρόβλημα. Νομίζω ότι έχουμε ήδη επιδείξει αρκετή ευελιξία, τον επάξει μεγαλύτερη ευελιξία εις βάρος της ε, πολιτικής συνοχής, δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσει από αυτού το Κοινοβούλιο. Και τελικά δεν ξέρω ποια είναι η χώρα εκείνη που θα ήταν πρόθυμη να παραιτηθεί μόνη της από τα κονδύλια συνοχής. Έχω την εντύπωση ότι το Κομισιόν, η Κομισιόν έτσι και αλλιώ δεν έχει την πρόθεση να περικόψει τα κονδύλια αυτά τουλάχιστον μέχρι το 2020. Αυτό που επίση με ενδιαφέρει είναι το χάσμα που υπάρχει στη χρηματοδότηση, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα να χρηματοδοτηθούν τα κενά μέχρι το τέλος αυτού του έτους. Αλλά ξέρετε, εγώ ε, πιστεύω ότι τελικά ε, αυτό είναι μόνο προσωρινή λύση του προβλήματος, γιατί ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι με την πολιτική συνοχή για διάφορους λόγους ξεκινήσαμε πολύ αργά και αυτή τη στιγμή δεν καταβάλλεται σχεδόν κανένα νέο πρόγραμμα για χρηματοδότηση. Άρα δηλαδή, όπως πάντα, περιμένουμε την, να ολοκληρωθεί η περίοδος χρηματοδότησης και μετά καταβάλλονται τα αιτήματα για χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη. Αν λοιπόν τα πράγματα συνεχιστούν με την πεπατημένη, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα όπως συνέβη και κατά την τελευταία περίοδο, ίσως και ακόμα ε, πιο ξημένο. Εσείς για την ενδιάμεση αναθεώρηση του ε, δημοσιονομικού πλαισίου έχετε κάποια ιδέα, έχετε κάποια πρόταση για να αντιμετωπιστεί αυτή η δυσκολία. Και τελευταίο μου ερώτημα την ε, ενδιάμεση αξιολόγηση τη συσχετίσατε μόνο με το ε, μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα. Εμείς όμως ε, χρειαζόμαστε και την μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής η Κομισιόν παρακαλώ πολύ μέχρι το τέλος του έτους ε, να υποβάλει προτάσεις άμεσα στο πλαίσιο της ε, πολιτικής συνοχής. Γιατί αν δούμε λιγάκι το χρονοδιάγραμμα, κοιτάξτε, το 19 θα έχουμε εκλογές, ε, ευρωπαϊκές εκλογές, άρα δηλαδή αν το 18 δεν έχουμε ολοκληρώσει ήδη τις διαπραγματεύσεις, τότε το 2020 δεν θα μπορεί να ξεκινήσει καμία νέα διαρθρωτική πολιτική. Προφανώς αυτό αφορά και άλλα μακροπρόθεσμα προγράμματα, άρα δηλαδή θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν η Κομισιόν να καταθέσει τις σχετικές προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, εκπρόσωποι του ECR δεν είναι παρόντες, ο λόγος του κύριο Γιάκοφτσιτς, εκ μέρους των φιλελευθέρων. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε που ήρθατε εδώ σήμερα και μας αφιερώνετε χρόνο. Είναι πολύ καλό να διατηρούμε τη συνέχεια των επαφών μας. Ακούσατε τους προηγούμενους ομιλητές συμφωνώ σε πολλά πράγματα μαζί τους. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί και να αναθεωρηθεί η πολιτική συνοχή. Δεν μπορούμε να την καταργήσουμε. Η πολιτική συνοχή αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι δεν είμαι σίγουρος ότι είναι βιώσιμη. Πρέπει να την προσαρμόσουμε τα επόμενα χρόνια και να την ευθυγραμμίσουμε με τις, πολιτικές, τις άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της συνέργειας ανάμεσα στο εύση και την πολιτική συνοχής. Είναι μεγάλη σημασία αυτή η συνέργεια, διότι πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η χρήση των κονδυλίων που διαθέτει η Κομισιόν μέσω του ΕΦΣΥ. Τώρα, ένα πρακτικό σχόλιο ως εισηγητής για την μακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιωνίου. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν και άλλες μακροπεριφέρειες της Βαλτικής. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε την αλπική υπερπεριφέρεια. Οπότε θα ήθελα να πω το εξής πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική συνοχή για τη χρηματοδότηση αυτών των μακροπεριφερειών. Γιατί οι στρατηγικές, οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές είναι πραγματικά έχουν αγγίξει τους πληθυσμούς. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική συνοχή για να τις χρηματοδοτήσουμε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται το Κοινοβούλιο να λάβει ε, θέση, αλλά μόνο αν χρηματοδοτηθούν οι μακροπεριφέρειες μπορούν να πείσουν. Και θα πρέπει να δείξουμε στους πολίτες ότι είμαστε κοντά τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ο κύριος Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγική σας παρέμβαση, η οποία μας επιτρέπει να κάνουμε συζήτηση επί της ουσίας για την περιφερειακή πολιτική και το μέλλον αυτής. Το είπατε και εσείς. Μιλούμε για 350 δις ευρώ, τα οποία στηρίζουν τις επιδιώξεις του χαρτοφυλακίου σας τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Και είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά αυτή και η περιφερειακή πολιτική έρχεται να μετριάσει στις περιφέρειες τις επιπτώσεις της κρίσης. Οφείλουμε όμως να μην ε, λησμονούμε τον βασικό στόχο της πολιτικής συνοχής που είναι η μόνη μεγάλη πολιτική αλληλεγγύης και ο στόχος της πολιτικής συνοχής είναι η μείωση των ανισοτήτων και των χασμάτων μεταξύ ε, των διαφόρων εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διαφόρων επικρατιών. Και όλα δείχνουν ότι παρά την προσπάθεια οι ανισότητες και οι αποκλήσεις όλο και οξύνονται. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό παρόλο που το γεωγραφικό κριτήριο δεν ελήφθη υπόψη για το ΕΦΣΥ, να παραμένει αυτή η μέρημνα, αυτό το μέλημα, γιατί η αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, αν δεν ληφθεί υπόψη το γεωγραφικό κριτήριο, θα συμβάλλει στην επιδίωξη στόχων που αντίκειται ε, στις συνθήκες. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερον, για την προσφυγική κρίση θα ήθελα να πω τα εξή. Η κρίση αυτή επιβαρύνει όλο το πρόγραμμα εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την πολιτική συνοχή, η οποία ε, σχετίζεται ε, θα πληγεί. Θεωρώ ότι μπορούμε να κινητοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία για να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Θέλω όμως να μοιραστώ μαζί σας μια ιδέα η οποία είναι δική μου και προσωπικώς είναι κάτι που με ανησυχεί. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων διαπραγματεύσεων ε, είχαμε προαπαιτούμενα και αιρεσιμότητα μακροοικονομικής φύσεως. Ξέρετε ότι πιστεύω ότι υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις σήμερα και εάν οι στόχοι π.χ. του ελλείμματος δεν τηρούνται, τότε υπάρχει ο κίνδυνος αναστολής του δικαιώματος αξιοποίηση των κονδυλίων για την εκάστοτε χώρα. Αυτό υπάρχει ήδη. Βλέπουμε όμως σήμερα πάρα πολλές χώρες μέλη να εποφελούνται και μάλιστα συνεχώς και επανειλημμένως ε, από τα διαρθρωτικά ταμεία και να μην σέβονται τις ευρωπαϊκές αξίες και να μην συμβάλλουν στην επιδίωξη λύσεων στο προσφυγικό. Και πέρα από τη κρίση την προσφυγική διαπιστώνονται και καταστρατηγήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ε, σε αυτό το πεδίο. Επομένως, Σήμερα που ο κίνδυνος για την Ευρώπη είναι θανάσιμος, ο κίνδυνος από τη μη τήρηση των αξιών που βρίσκονται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών συνθήκων. Σήμερα λοιπόν με όλα αυτά τα δεδομένα οφείλουμε να προβληματιστούμε για διαδικασίες κυρώσεων ή προαπαιτουμένων αν θέλετε για τις χώρες που δεν σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, για τις χώρες που δεν σέβονται τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι η εξής. Έχει να κάνει με μια πρόταση που κατατέθηκε πρόσφατα από το Ίδρυμα Jacques Delors. Ε, το πρόταση που μας καλεί να αναδιατυπώσουμε τη ρήτρα των προβλεπόμενων επενδύσεων στο Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας. Γνωρίζετε ότι ιδιαίτερος στη ζώνη του ευρώ οι χώρες που χρειάζονται περισσότερο ευελιξία σήμερα στερούνται τις δυνατότητες να να αξιοποιήσουν αυτή τη ρήτρα. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω σε μία πρόταση η οποία θα επιτρέψει σε ορισμένες χώρες που χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις σήμερα να μπορέσουν οι χώρες αυτές να αξιοποιήσουν αυτή τη ρήτρα, να ωφεληθούν από αυτή χωρίς να ελοχεύει ο κίνδυνος να υπαχθούν σε ε, διαδικασίες ε, ε, διάφορες και γνωστές. Σε κάθε περίπτωση, πριν από δύο εβδομάδες ήμουν στη διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκουσα τις δεσμεύσεις σας, ήταν εκεί παρόν και ελπίζω τα έργα που θα υποβληθούν από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες να είναι επιλέξιμα υμφίνε των αιώνα τον άπαντα. Είπατε ότι η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική και εμείς έχουμε κάνει αυτό το ε, αυτή τη δουλειά στις από κέντρους περιφέρειες. Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από το να καταρρεύσουν οι ελπίδες μας. Ευχαριστώ κύριε Βάνα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω που ε, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Πάρα πολλά αυτά είπατε, ήδη αναφέρθηκαν από τους ε, προλαλήσαντες. Εγώ να εστιάσω την προσοχή μου σε δύο συγκεκριμένα ερωτήματα που και τα δύο αφορούν το Στρατηγικό Ταμείο Επενδύσεων και τους ε, στόχους του. Αφορούν και στην σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, ε, το βιώσιμο πρόγραμμα για ενεργειακά θέματα και εκεί αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην πυρηνική ενέργεια. Ξέρετε, εγώ προέρχομαι από τους ε, πράσινους και θέλω να σας πω ότι ήδη όταν συστήθηκε αυτό το ταμείο εμείς ε, είχαμε την, το φόβο ότι ειδικά στην περίπτωση αυτή το μόνο ο μόνος στόχος θα μπορούσε να είναι η στήριξη της πυρηνικής ενέργειας η αναγέννηση της πυρηνικής ενέργειας, επιτρέψτε μου να πω. Εγώ έρχομαι από την Αυστρία και βεβαίως ε, το θέμα της πυρηνικής ενέργειας πρέπει να σας πω ότι είναι ένα θέμα που ευαισθητοποιεί όλα τα κόμματα και οι πολίτες κρίναν ότι είναι μεγάλη επιτυχία για μας ε, το ότι είχαμε αποκλείσει την ε, χρηματοδότηση πυρηνικής ενέργειας στην Αυστρία από αυτό το νέο ταμείο. Εσείς λοιπόν με αυτό το έγγραφο που καταρτήσατε, εκεί ε, ορίζεται ως χρηματοδότες όχι μόνο το ΕΦΣΥ αλλά και την πολιτική συνοχής για την πυρηνική ενέργεια. Τι ακριβώς συμβαίνει. Και ένα δεύτερο ερώτημα για το ΕΦΣΥ. Πρόκειται για το εξής. Όσον αφορά τους κανόνες του ΕΦΣΙ, αναφέρεται με απόλυτη σαφήνεια ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει προστασία για, για μια συγκεκριμένη επένδυση, στην περίπτωση αυτή, μια δόση που δεν καταβάλλεται θα πρέπει να αναλαμβάνεται από το Ταμείο Επενδύσεων. Σε περίπτωση μη καταβολής δηλαδή μια δόση από το ΕΦΣΥ, τη δόση αυτή την αναλαμβάνει να την καταβάλει το Ταμείο Επενδύσεων. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε ε, πώς είναι δυνατόν να λυθεί αυτή η αντίφαση και κυρίως όσον αφορά το θέμα της ε, νομικής ασφάλειας ε, κατά την χρήση των κονδυλίων. Ντεμάτο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καλωσορίσατε. Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι οι επενδύσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτω του 15% σε σχέση με το επίπεδο προ-κρίσης. Άρα δηλαδή αυτή η συνταγή της ε, ε, λιτότητας οδήγησε σε χειρότερη κατάσταση του ασθενού. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε το Διαρθρωτικό Ταμείο που κάνει επενδύσεις και αυτό αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, ε, αφορά και θέμα συνοχής. Το δεύτερο, το εψ ε, αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί τι θα κάνει. Πέρα από το γρίφο ε, σχετικά με το πολλαπλασιαστή για τις ιδιωτικές επενδύσεις, εμείς περιμένουμε ακόμα τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία σχετικά με τη μόχλευση. Προβλέπονται εγγυήσει για θέματα ενέργειας, για την ε, χρήση του ε, αερίου. Αυτά όμως ενισχύουν όλα τις μεγάλες επιχειρήσεις, όπως ε, στην περίπτωση των μονάδων για το φυσικό αέριο, σαν παράδειγμα το αναφέρω αυτό. Υπάρχουν επίσης ε, και διάφορες άλλες ε, λεπτομέρειες ε, σχετικά με τα κονδύλια που τα χορηγούνται σε συγκεκριμένες μονάδες των κρατών μελών. Υπάρχει ένας τεράστιος λαβύρινθος δηλαδή των δημόσιων και των ιδιωτικών κονδυλίων. Εμείς θα θέλαμε να ενημερωθούμε περισσότερο γι' αυτό. Ας πούμε ένα πρόγραμμα περίεργο, Ιρλανδικό, Renewable Income Europe, ένα πρόγραμμα που το προωθεί η BlackRock στην Ελλάδα το ξέρουν αυτό πάρα πολύ καλά, γιατί ενεπλάκη και η Ελληνική Τράπεζα στο τραπεζικό σύστημα του 2011. Υπάρχουν λοιπόν πολλά που έχουν σχέση και με τις ε, εγγύησει ε, που πρέπει να δίδονται στην περίπτωση της BlackRock όμως ε, δεν αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία αυτά και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη διαφάνειας. Τέλος, για να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα στο θέμα της συμπληρωματικότητας σχετικά με τα κονδύλια που δίδονται για επενδύσεις και το ΕΦΣΥ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι υπάρχουν κονδύλια τα οποία αφαιρούνται από τη συνοχή και από τον ορίζοντα 2020 και αυτά για να φαίνεται πολύ πιο μεγάλο το πρόγραμμα Juncker. Άρα δηλαδή υπάρχουν δύο διαφορετικές ε, δύο διαφορετικοί θεσμοί που παρότι υποτίθεται ότι είναι συμπληρωματικοί τελικά δημιουργούν σύγχυση κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτά όλα αποβαίνουν εις βάρος των περιφερειακών και των τοπικών πολιτικών. Πολύ ωραία. Αυτές ήταν ερωτήσεις από τους συντονιστές. Άλλους ε, τρεις, πέντε έχω που έχουν ζητήσει το λόγο. Έξι τελικά. Εντάξει, σας είδαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα σας ήθελα να δώσετε τώρα το λόγο για να απαντήσετε και μετά θα συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Thank you very much. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις. Πρώτον, για το FC. Σας δώσω μερικά νούμερα. Γράψτε τα. 64 επενδυτικά σχέδια έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί. Ή μηχανικές επενδύσεις ή επενδύσεις σε υποδομές. 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση αυτών των 64 έργων. Επιπλέον, 185 συμφωνίες έχουν συναφθεί με ενδιάμεσες τράπεζες για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται μέσω τραπεζών. 3,5 δισεκατομμύρια τα κονδύλια για αυτές τις χρηματοδοτήσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 185 λοιπόν τράπεζες έχουν συμφωνήσει μαζί μας και θα χρηματοδοτήσουν 142.000 ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 142.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν μέσω των 185 τραπεζών με τις οποίες έχουμε υπογράψει συμφωνίες. Αν προσθέσουμε την χρηματοδότηση του ΕΦΣΙ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα μεγαλύτερα έργα, έχουμε ένα σύνολο 12 και κάτι δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι το οποίο θα μοχλεύσει 100, πάνω από 100 δισεκατομμύρια από τον ιδιωτικό τομέα. Όταν δημιουργήθηκε αυτό το ταμείο, κάποιοι λέγανε ότι είναι μαγεία και ότι δεν πρόκειται να ε, μαζευτούν αυτά τα χρήματα. Όμως, 140.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα έχουν δει τα χρήματα αυτά με χρήση 12 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον Ευρωπαίο Φορολογούμενο μοχλεύσαμε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ιδιωτικών κεφαλαίων. Είμαστε διαφανείς, ενημερώνουμε και ε, προσπαθούμε έτσι ώστε όλες οι περιφέρειες, όλες οι χώρες, όλες οι επιχείρησεις να μπορούν να τα αντιγράψουν αυτά αν υπάρχει κάποιος που δεν με ακολουθεί στο Twitter, δεν με διαβάζει στο Twitter, ε, σας ενθαρρύνω να το κάνει, τον να το κάνει. Γιατί ενημερώνω τακτικά και λεπτομερώς και μπορείτε να βρείτε και πολύ καλά παραδείγματα για να αντιγράψετε. Το ΕΦΣΙ λειτουργεί αρκετά καλά. Ένα από τα προβλήματα είναι η έλλειψη γνώσης, συνειδητοποίησης ευαισθητοποίηση, διότι δεν γνωρίζουν οι πάντε το τι έχουμε να προσφέρουμε και εκεί χρειάζομαι τη βοήθειά σα. Θα είμαι και πάλι ειλικρινή. Ε, γνωρίζω ελάχιστου ευρωβουλευτέ που έχουν κάνει κάτι για να διαδώσουν το ΕΦΣΥ. Ελάχιστου. Εσεί είσαστε πολύ όμω και γνωρίζετε τι μπορεί να κάνει το ΕΦΣΥ. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να περάσετε το μήνυμα για το τι έκανε ήδη το ΕΦΣΥ. Αν χρειάζεστε περισσότερη τεκμηρίωση, μπορούμε να σας δώσουμε ό,τι χρειάζεστε. Όλα τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται θα τα βρείτε στο site. Πολύ καινοτόμα έργα. Για παράδειγμα, η πλατφόρμα απο... ενεργειακής αποδοτικότητας. 40.000 οι κατοικίες στη Γαλλία. Ε, έχουν χρηματοδοτηθεί για να ανακαινιστούν ενεργειακά. Αυτό το παράδειγμα μπορεί να αντιγραφεί και σε άλλες περιοχές. Μετά, πάρτε έναν ευρωβουλευτή από την Πορτογαλία, για παράδειγμα, ή από την Κύπρο. Θα καλούσαν στι στη του επιχειρηματίε, τράπεζε, εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην χώρα του, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο κλπ. και έναν εκπρόσωπο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όλοι αυτοί μαζί θα μπορούσαν ε, να συζητήσουν πώς θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα, για παράδειγμα, του ε, αναγέννησης ε, καταλημά, τουριστικών καταλημάτων. Χιλιάδες επιχειρηματίες οι οποίοι δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν με λογικούς ε, όρους για την ενεργειακή ε, ανακαίνιση των κτηρίων τους, θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν μέσω μιας τέτοιας πλατφόρμας η χρηματοδότηση θα μπορούσε να γίνει με πολύ πιο οικονομικούς όρους και ενδεχομένως θα ήταν και ο μόνος τρόπος. Οπότε ε, το ΕΦΣΙ τι κάνει, ε, ματσάρει, ε, ζευγαρώνει τις ανάγκες με του, τη χρηματοδότηση. Κύριε Σπυράκη είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ευρωβουλευτού που έχει κάνει πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Ε, αν πουλήσετε δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στους επιχειρηματίες σας, εμείς δεν πρέπει να πάρουμε προμήθεια, αλλά είναι ωφέλιμο, διότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται θέσεις εργασία και ρέει χρήμα. Είναι στη διάθεσή σας, όσο και στη δική μας. Οπότε συνεργαστούμε στενά. Κύριε Κρέιλ, κύριε Κρέιλ, ε, ρώτησε για την πολιτική συνοχή και το κατά πόσο είναι απερχιωμένη. Όχι απαραίτητα, αλλά σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί. Ε, τα χρηματοδοτικά μέσα και οι επιδοτήσεις ε, αυτή τη στιγμή η χρηματοδότηση θα παραμείνει εστιασμένη στις επιδοτήσεις, αλλά σίγουρα θα έπρεπε να σκεφτούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα χρηματοδοτικά μέσα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για παράδειγμα, είναι ε, σημαντικοί δικαιούχοι τέτοιας βοήθειας ε, και μπορούμε να συνδυάσουμε τα διαφορετικά ταμεία μαζί με το ΕΦΣΥ. Μάλιστα είχαμε ε, ε, ε, θέλουμε να δημοσιεύσουμε μια ανακοίνωση για αυτό το θέμα, αλλά οι κανόνε είναι περίπλοκοι. Ξέρουμε πώς μπορεί να γίνει, αλλά είναι περίπλοκο. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε τις, ένα hub της υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις επενδύσεις στην Ευρώπη. προκειμένου να βοηθήσουμε τις περιφέρειες ή τα κράτη-μέλη να συνδυάσουν το ΕΦΣΥ με τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Αν έχετε πληροφορίες εσεί οι ίδιοι για τέτοιε προσπάθειες, ενημερώστε μας αυτό το, το hub, αυτέ οι συμβουλευτικές υπηρεσίε που έχουμε, η συμβουλευτική υπηρεσία που έχουμε δημιουργήσει, ε, μπορούν να σας συμβουλεύσουν για το πώ μπορεί να δημιουργηθεί μια επενδυτική πλατφόρμα ή να χρησιμοποιηθούν από κοινού το ΕΦΣΙ και τα διαρθρωτικά ταμεία. Ε, μακροοικονομικές αρισιμότητε. Ε, ας δούμε την πραγματικότητα. Αν μια κυβέρνηση για οποιοδήποτε λόγο ιστερεί στην ε, δημόσια χρηματοδότηση, αυτό συνήθως οδηγεί σε φτωχοποίηση. Αν όμως η ίδια χώρα υπόσχεται και αποφασίζει να ε, μεταρρυθμίσει την πολιτική της, γιατί ο κόσμος αλλάζει, αυτό δεν έχει σχέση με το έλλειμμα ή με το χρέος και μπορεί να βοηθηθεί. Χρησιμοποιούμε τα χρήματα των φορολογουμένων και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες να έχουν σε τάξη τα οικονομικά τους, τα δημοσιονομικά τους. Αν δούμε και άλλες πολιτικές εκτός της οικονομικής πολιτικής. Αν, κάποια χώρα σκοπίμως παραβιάζει το κράτος δικαίου. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτή τη χώρα δίνοντας χρήματα στην κυβέρνησή της. Είμαστε και μια ένωση αρχών και αξιών. Οπότε οι πόροι μας θα πρέπει να δαπανώνται σύμφωνα με αυτές τις αρχές. Τώρα, ενθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Δεν είμαι ειδικό. Η Κρυσταλίνα Γκεργίεβα, η συνάδελφός μου, ε, γνωρίζει καλύτερα την κατάσταση. δεν νομίζω ότι κάποιος έχει πει πως ε, θέλει να πληρώνει παραπάνω ή θέλει να πληρώνει για τους άλλους, για να πληρώνει λιγότερο. Μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά στην καλύτερη περίπτωση πιστεύω ότι ε, θα καταφέρουμε να δαπανούμε με καλύτερο τρόπο χρήματα τα οποία ήδη έχουμε. Ναι, αυτό που είπατε είναι και αυτό μια εναλλακτική λύση. Χρήματα τα οποία ε, έχουν περισσέψει να μην επιστρέφονται στα κράτη-μέλη αλλά να επαναχρησιμοποιούνται. Με λίγο, δηλαδή να τα δαπανούμε με λίγο διαφορετικό τρόπο έτσι ώστε να βελτιώνουν τα αποτελέσματα. Η Κρυσταλίνα Γεωργίβα είναι υπεύθυνη για τον προπολογισμό. Ε, θα πρέπει να το δούμε. Τώρα, το αν το ΕΦΣΥ θα, η προγραμματική περίοδος θα φέρει σημαντικές αλλαγές στα κράτη που είναι κάτω του μεσουόρου. Οικονομικά εννοώ. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα την πραγματικότητα. Να κάνω όμως ένα σχόλιο η... θα πρέπει να ακούσουμε τις συμβουλευτικές υπηρεσίε. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να αυξηθεί η απορροφητικότητα. Και μόνο έτσι μπορούμε να επωφεληθούμε στα μέγιστα του ΕΦΣΥ. Υπάρχουν έργα του ΕΦΣΥ σε 26 κράτη-μέλη. Μόνο η Μάλτα και η Κύπρος δεν έχουν ακόμα κάποιο έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΦΣΥ. Εργαζόμαστε όμως και με αυτές τις χώρες. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο οι διοικητικές ελλείψεις. Πάρτε τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Στη Βουλγαρία οι ιδιωτικές τράπεζες είναι πάρα πολύ δραστήριες στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, εκεί δεν χρειάζεται να εμπλακούν ιδιαίτερα οι κρατικές αρχές. Οι οι τράπεζε αντλούν χρήματα από τον ΕΦΣΥ. Αυτό δεν σημαίνει στη Ρουμανία από την άλλη μεριά. Εργαζόμαστε σε αυτό το θέμα όμω. Αλλά θα πρέπει να ακούσουμε τι μας λένε οι βουλευτικέ υπηρεσίε προκειμένου όλες οι χώρες να επωφεληθούν εξίσου. Πυρηνική ενέργεια και εύση. Το εύση δεν έχει χρηματοδοτήσει ούτε και θα χρηματοδοτήσει η πυρηνική ενέργεια ο κλάδος ο οποίος πιο πολύ έχει χρησιμοποιήσει ε, χρήματα από τον ΕΦΣΥ είναι η, ενεργειακή αποδοτικότητα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί εκεί είναι το μέλλον. Και ο ΕΦΣΥ προσπαθεί να καλύψει τα κοινά του ιδιωτικού τομέα όταν ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι πρόθυμος να χρηματοδοτήσει νέες τεχνολογίες για την ενεργειακή απόδοση ή για τις με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα παράδειγμα που ελπίζω να μην το έχω πει πιο παλιότερα είναι το εξής. Στη Δανία ε, έχω κάνει το εξής που μπορεί να αντιγραφεί. Δημιούργησαν ένα ιδιωτικό επενδυτικό ταμείο προς το οποίο, ε, του οποίου ε, το ΕΦΣΙ αγόρασε μετοχές και είναι αυτό το οποίο θα καλύψει οποιαδήποτε, οποιαδήποτε προκύψουν. Ε, το, το συνολικό ταμείο είναι, έχει κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων και αυτό το ιδιωτικό πνευματικό ταμείο της Δανίας θα χρηματοδοτήσει έργα ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Βόρεια Ευρώπη και χρηματοδοτείται από ε, ταμεία, από τα κεφάλαια συνταξιωτικών ταμείων. Και από τον ΕΦΣΙ βέβαια. Αυτό το μοντέλο μπορεί να αντιγραφεί και αλλού. Συνταξιδοτικά ταμεία τα οποία χρηματοδοτούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, χρηματοδοτούν την καινοτομία. Uh, Ε, η τι θα γινόταν αν η, ε, δεν είχε γίνει ε, δημοσιονομική ε, εξυγίανση. Θα ήταν χειρότερη η κατάσταση. Βέβαια έχουμε ήδη λιγότερες επενδύσεις, αλλά θα ήταν ακόμα λιγότερη. αυτή τη στιγμή όμως ε, αυξάνονται οι κρατικές επενδύσεις. Ε, και ακόμα δεν έχουμε δει όλο, όλη την, το, το όφελος προκύπτει από τον ΕΦΣΥ. Οι επενδύσεις θα επανέλθουν όταν οι επενδυτές ε, ξανιώσουν εμπιστοσύνη στο μέλλον της χώρας, κάθε χώρας. Οπότε η δημοσιονομική πολιτική είναι σημαντική για τη βελτίωση αυτής της ε, κατάστασης για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για την αύξηση των επενδύσεων. Okay. Yeah. One maybe additional uh, aspect to renewable energies and... Τώρα για τη βιομάζα μεταξύ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ήδη το ΕΦΣΥ χρηματοδοτεί σχέδια, έργα που εμπλέκουν τη βιομάζα. Η βιομάζα χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο πλέον. Ε, για παράδειγμα είναι εργοστάσια τα οποία εξυγχρονίζονται έτσι ώστε να χρησιμοποιούν το 100% της βιομάζας. Για παράδειγμα, το ευσύ χρηματοδοτεί έργα τα οποία ε, αποσκοπούν στο να παραχθούν υποπροϊόντα από τη χρήση βιομάζας. Ε, βιοπροϊόντα, ε, ε, υποπροϊόντα. Θα πρέπει όμως να αντιγράψετε παραδείγματα από το site μας να βοηθήσετε τις, περιοχές, τις περιφέρειες της χώρας σας να εκμεταλλευτούν πλήρως το ΕΦΣΥ. Και μπορούμε να σας βοηθήσουμε ό,τι χρειάζεται. I asked, uh, uh, the development of... Ως προς ε, την κατάληξη, την κατάσταση με την ε, ε, απόσταση μεταξύ πληρωμών και ετοιμάτων πληρωμής με την απόκληση μεταξύ των δύο. Θα κάνετε κάτι, είπατε ότι θα επιταχυνθεί αυτό κατά τη διάρκεια του 2016. Απάντηση. Καλύτερα να απαντήσει στην ερώτηση αυτή η συνάδελφος Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, γιατί είναι πιο εξοικειωμένη με το ζήτημα. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να απευθύνουμε το ερώτημα στην κυρία Γεωργίευα τον Ιούλιο που θα τη δούμε. Έξι ομιλητέ που θα πάρουν το λόγο. Θα ήθελα να μην ξεπεράσει ο καθένας τα δύο λεπτά για να μπορέσει και ο κύριος Κατάινεν να απαντήσει. Η κυρία Μάλετιτς παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχω ένα ερώτημα για τις συνέργειες μεταξύ του ΕΦΣΙ και του ΕΣΥΦ. Όταν ε, αν δούμε τα project, τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό Ταμείο και το Επενδυτικό Ταμείο, έχουμε συγχρηματοδότηση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει συγχρηματοδότηση όχι μόνο για το εθνικό σκέλος αλλά και για το μη επιλέξιμο σκέλος της χρηματοδότησης. Τώρα, εάν δούμε τα έργα των ιδιωτών που μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης από το ΕΣΥΦ, έχουμε τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις όπως γνωρίζετε και Βάσει των κανόνων αυτών δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει άλλους πόρους όπως είναι το ΕΦΣΥ. Και από εκεί και πέρα έχουμε και γενικότερους κανόνες που είναι σε ισχύ. Διαφορετικό υλικό τεκμηρίωσης για το φάκελο υποψηφιότητας επιλεξιμότητας για το ΕΦΣΙ και διαφορετικό για το ΕΣΥΦ. Αλλά και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής είναι διαφορετικά. Πώς θα έχουμε συνέργεια με τόσες διαφορές τελικά. Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται κατά την άποψή μου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα, για το ότι μας ενθαρρύνεται να διαδώσουμε αυτό το μήνυμα στις χώρες μας, ότι μπορούν περισσότερο οι περιφερείς να αξιοποιήσουν τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και θα πρέπει να απευθυνθούμε και στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί και αυτές μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα κονδύλια. Και παρόλο που γνωρίζω ότι έχετε επισκεφθεί πολλά κράτη-μέλη, όταν οργανώνουμε κάποια διάσκεψη, κάποιο συνέδριο, ίσως μπορεί να έρθει κάποιος από τη γενική σας διεύθυνση, αν ναι, όχι εσείς, για να μας εξηγήσουν για τις διάφορες δυνατότητες. Ευχαριστώ ο κύριος Βόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο, διότι ήρθε ξανά να μας επευθύνει το λόγο. Ξέρετε, την πρώτη φορά που ήρθατε εδώ, καταστήσατε σαφές ότι δεν θα υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ ΕΦΣΥ και διαρθρωτικών ταμείων. Θέλετε τα καλύτερα project να χρηματοδοτούνται από το Σήμερα όμως λέτε ότι υπάρχουν ευκαιρίες να συνδυαστεί το ΕΦΣΙ με τα διαρθρωτικά ταμεία. Είναι χρήσιμο για μας να μας δώσετε κάποια παραδείγματα. Παραδείγματα που έχει αυτό συμβεί και πώς. Από εκεί και πέρα, ε, ζητήσατε και πληροφορίες. Είπατε ότι υπάρχει μια συμβουλευτική υπηρεσία διαθέσιμη. Μπορείτε να το αναπτύξετε αυτό το θέμα. Ποιος είναι ο ρόλος αυτής της ε, συμβουλευτικής υπηρεσίας. Και δεύτερη παρατήρηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εγώ είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Βλέπετε ότι και καταλαβαίνετε ότι δεν έχω καμία πρεμούρα να δω τις προτάσεις σας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είμαι διατεθειμένος να περιμένω, να έρθουν. Ε, ίσως να έχουμε αύξηση των πληρωμών στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Μιλήσατε για την ευελιξία. Και αυτό είναι σημαντικό. Να δούμε και το θέμα της καθυστέρησης των πληρωμών. Φαίνεται τεχνική αυτή για τεχνικούς λόγους, όμως αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους δικαιούχους όταν δεν υπάρχει ροή στην πληρωμή των δαπανών τους. Και τέλος, το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Αναφέρθηκε και η Κωνσταντς Κρέλ σε αυτό. Ε, είναι κάτι το πολύ σημαντικό και από την οικονομική σκοπιά και από τη δημοσιονομική, χρηματοδοτική και χρηματοπιστωτική σκοπιά για τις περιφέρειες. Αλλά και το πολιτικό μήνυμα είναι τεράστιο και πολύ σημαντικό για πάρα πολλούς ανθρώπους το να υπάρχει μια ποινική που να δείχνει ότι το έργο εν μέρη πράγματι χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και ο μόνος λόγος που οι άνθρωποι την επιθυμούν. Πρέπει δηλαδή να έχουμε ένα σύστημα που να βασίζεται στα αποτελέσματα, οι επιδόσεις να μετρώνται με τα αποτελέσματα. Δεν θέλουμε αυτό να είναι δικαιολογία για να αποκλείονται οι περιφέρειες και δεν θέλουμε αυτόματες κυρώσεις και πέναλτι για έργα που δεν ευωδώνονται. Το σημαντικό είναι να μπορούμε να δείξουμε στο μέλλον ότι ε, Εάν θέλουμε να προστατεύσουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τα κονδύλια για τις περιφέρειες, θα πρέπει να μπορούμε να δείξουμε ότι είναι αποτελεσματικά, δουλεύουν και φέρνουν αποτελέσματα. Έχετε ιδέες γι' αυτό, δηλαδή να έχουμε προϋπολογισμό που να καταρτίζεται με βάση τις επιδόσεις. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Ροντρίγκης, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ τον Επιτρόπο για την παρουσία του. Δεν θα σχολιάσω την παρέμβαση της ε, Κομισιόν στην, ε, στον πορτογαλικό τραπεζικό τομέα, όπως για παράδειγμα στην Πανίφ ε, και με τα τραγικές συνέπειες που είχε στην Μαδέρα, στην περιφέρεια μου. Ξέρω ότι εσείς είσαστε ιδιαίτερα ευαίσθητος για το θέμα των ε, ακρός περιφερειακών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εξόχως των περιοχών είναι περιοχές οι οποίες έχουν σημαντικά προβλήματα. Οπότε οι ερωτήσεις μου ε, είναι εξή. Πρόκειται για περιοχές οι οποίες πληθώνται ιδιαίτερα από την μετανάστευση, από την απασχόληση. Ε, μετανάστευση εννοώ ότι τις εγκαταλείπει ο πληθυσμός τους πιο πολύ. Ε, σε ό,τι αφορά την ανεργία ε, ε, είναι ψηλή και ταυτόχρονα δεν έχουμε επαγγελματική κινητικότητα όπως αναφέρεται, αλλά πραγματικά μετανάστευση για καλύτερη τύχη. Πώς μιλάμε για ανταγωνιστικότητα όταν μερικές από αυτές τις περιοχές ε, έχουν πρόσβαση στην υπηρετική Ευρώπη μόνο μέσω αεροπλάνου. Οπότε η μεταφορά αγαθών είναι πραγματικά πολύ ακριβή. Μετά, ε, έρευνα και καινοτομία. Οι ερευνητές ε, είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσει κανείς ένα ισχυρό ερευνητικό κέντρο σε αυτές τις περιοχές. Τι λοιπόν πέραν του άρθρου 349 υπάρχει ως κίνητρο για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα. Ποια ε, θετική διάκριση στον τομέα των μεταφορών για παράδειγμα. Το, το, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για παράδειγμα, δεν έχει φτάσει καλά-καλά στη Μαδέρα. Η κεντρική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη. Ε, και ε, μας παραπέμπει στην Ευρώπη και η Κομισιό μας παραπέμπει στην ε, κυβέρνησή μας. Μετά, ε, ως αντιπρόεδρος της Euromed ε, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα το θέμα των προσφύγων. πρέπει ιδιαίτερα να αναθεωρηθεί η συμφωνία και το πρόγραμμα με την Τουρκία. Δεν συμφωνώ να πούμε ότι η πολιτική συνοχής ε, κρίνεται με βάση τα αποτελέσματα. Ε, μην ξεχνάμε ότι κάθε περιοχή ξεκινάει από διαφορετική αφετηρία. Οπότε δεν μπορούμε να ε, συγκρίνουμε τα τελικά αποτελέσματα μόνο. θα πρέπει ε, να ληφθούν διαστοτικά μέτρα για αυτές τις περιοχές. Τέλος, για την μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Αυτές οι περιοχές έχουν, πρέπει να έχουν διοικητική και οικονομική αυτονομία. Οι Αζόρες ε, πάντοτε τηρούσε το κριτήριο του ελλείμματος, η Μαδέρα όχι. Παρ' όλα αυτά, καμία από τις δύο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια. Δεν είναι άδικο. Ε, γιατί δεν χρησιμοποιούμε άλλα κριτήρια που έχουν πιο πολύ σχέση με τον άνθρωπο. Ευχαριστώ κύριε Σπυράκη. Σα Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ε, για όλα τα κύριε Επίτροπε για τα πολύ καλά σας λόγια. Κοιτάξτε, όσον αφορά τη συμπληρωματικότητα των δύο ταμείων, του ΕΣΥΤ και του ΕΦΣΥ, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει και έλλειψη ε, διαχείρισης και απορρόφησης κοντιλίων σε πολλά κράτη-μέλη. Και ως παράδειγμα θα μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία από την Ελλάδα με βάση την, μια τελευταία έκθεση που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στην Επιτροπή από πέντε δις των ε, λειτουργικών ε, περιφερειακών προγραμμάτων μόνο το 0,49% απορροφήθηκε. Επίσης, 13,4 δις ευρώ από τα ε, προγράμματα και από αυτά μόνο το 1,63 απορροφήθηκε. Άρα δηλαδή είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και θέλω να σας ρωτήσω ε, προβλέπετε κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για να ενθαρρύνετε τα κράτη-μέλη ε, προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης ε, απορροφητικότητας των κονδυλίων και μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι η χρήση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Ενταρρύνεται τα κράτη-μέλη να εξετάσουν και μια δεύτερη ματιά στο χαρτοφυλάκιό τους. Έχετε λοιπόν ίσω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Γνωρίζω ότι η Ιταλία έχει αναλάβει πρωτοβουλία σχετικά με τη χρηματοδότηση ε, από το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και ρωτώ από την Ελλάδα έχετε πάρει κάποιο αίτημα σχετικά ή όχι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς θέλετε να γίνει πιο γνωστό το ΕΦΣΥ. Εντάξει, συμφωνώ κι εγώ. Αλλά να πω όμως το εξή. Για να είναι κάτι γνωστό, να το διαδώσει κανεί, πρέπει καταρχήν να έχει πιστεί. Και θέλω λοιπόν να σας πω ότι οι έρευνες οι δικές μας, αλλά και αυτό το πολύ συγκεκριμένο που μας προτείνατε εσείς σήμερα, Εμένα τουλάχιστον δεν με έπεισαν για την αποτελεσματικότητά τους. Έχουμε τα προγράμματα ΕΦΣΙ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τα είδαμε λιγάκι, και στα προγράμματα που απαριθμούνται, δύο αφορούν ευρωπαϊκά κράτη. Μόνο δύο. Έχουμε λοιπόν την εντύπωση ότι η χρήση του ε, προγράμματος ΕΦΣΙ είναι άμεσα συνδεδεμένη με μεγάλα project, μεγάλα έργα. Αυτά αφορά και τη Γερμανία. Γι' αυτό λοιπόν έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση προς εσάς. Ειλικρινά πιστεύετε ότι αυτό το ταμείο το ΕΦΣΙ θα ωφελήσει εκείνες τις περιοχές όπου οι επενδύσεις είναι πολύ περιορισμένες. Δηλαδή πιστεύετε ότι αυτό το ταμείο θα καλύψει το κενό επενδύσεων που υπάρχει. Γιατί εγώ θέλω να σας πω ότι από τα στοιχεία που έχουμε τουλάχιστον εμείς δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Και ένα τρίτο ερώτημα. Θα ήθελα να γνωρίζω, να μας πείτε, αυτό που λέω τώρα έχει σχέση και με τα προηγούμενα, να γνωρίζω λοιπόν, όσον αφορά τη χρήση του ΕΦΣΙ στην Ελλάδα, να σας πω ότι από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία, μόνο ένα πρόγραμμα αφορά την Ελλάδα. Άρα δηλαδή ερωτώ, στοχεύεται στη στήριξη και πραγματοποίηση επενδύσεων που δεν έχουν γίνει ακόμα. Δηλαδή, θέλετε να κάνετε επενδύσεις, ναι ή όχι. Η τελευταία ερώτηση, Μανσκούρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, διότι ήλθατε για να μας μιλήσετε για το Ταμείο Συνοχής για την Περιφερειακή Πολιτική, μεταξύ άλλων. Να σας πω ότι προέρχομαι κι εγώ από μια εξόχως απόκεντρη περιφέρεια και, και προσυπογράφω απολύτως τα λόγια της συναδέλφου Ροντρίκες. Είπατε ότι οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες δεν γνωρίζουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν ε, από πλευράς χρηματοδότησης, κονδυλίων κτλ και μας καλέσατε να μεταβούμε επί τόπου και να διαδώσουμε αυτό το μήνυμα. Εγώ σας λέω ότι το κάνουμε. Εγώ προσωπικώς το κάνω συνεχώς. Γνωρίζω τις δυσκολίες που έχουμε γιατί είμαστε νησιωτική περιοχή. Όμως, θέλω να σας πω το εξής. Πολλής λόγος γίνεται για το μέλλον, το τι μέλη γενέστε με το Ταμείο Συνοχής μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε σήμερα. Υπάρχουν ανησυχίες. Θα, συνεχιστούν, θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά τα κονδύλια σε αυτά τα ταμεία, στο Ταμείο Συνοχής, γιατί στους διαδρόμους πολλά λέγονται. Για μένα αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ιδρυτικών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τίθεται στην υπηρεσία της αλληλεγγύης, η οποία δεν είναι μία λέξη άνευ νοήματος ειδικά, ειδικά για μας τους νησιώτες. Σε τι χρησιμεύει όλη αυτή η συζήτηση, όλη αυτή η παρέμβαση, αν δεν υπάρχουν εγγυήσει ότι αύριο και μεθαύριο, σε ένα ε, εγγύης και απότερο μέλλον, θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά τα ταμεία. Μπορείτε να διασκεδάσετε τις αμφιβολίες μας. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να παρέμβω κι εγώ ως μέλος της Επιτροπής ε, Περιφέρειας. Δεν θα θέσω ερωτήσεις, έχετε ήδη θέσει εσείς. Και θα λάβουμε απαντήσεις στο εγγύς μέλλον, ίσως. Θέλω όμως να δηλώσω ότι γνωρίζω πολύ καλά ότι η συνέργεια μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών ταμείων είναι κάτι το πολύ δημοφιλές στη Βουλγαρία. Εγώ θα εργαστώ προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω ότι μπορώ να βασίζομαι στη δική σας βοήθεια, στη βοήθεια του γραφείου σας, κύριε Αντιπρόεδρε. Μετά από αυτή τη δήλωση ε, θα σας δώσουμε την ευκαιρία να απαντήσετε για δεύτερη φορά. Ο Αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Για τη συμβουλευτική υπηρεσία καταρχάς να πω, όλα θα τα βρείτε στη διαδικτυακή πλατφόρμα του EAH, European Advisory Hub, στον Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Κόμβο. Έχουμε συγκεντρώσει εκεί την εμπειρογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και εκεί υπάρχει το email και το τηλέφωνο του αρμοδίου αναλόγως με την ερώτησή σας. Δεν ξέρω πόσες επαφές έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα, ε, περίπου 150. Και το 70% αυτών προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι μία δυνατότητα που προσφέρει ε, ε συμβουλές και ε, τεχνική βοήθεια και στον ιδιωτικό τομέα και στις δημόσιες αρχές, στη δημόσια διοίκηση, για όλα αυτά τα θέματα. Και αυτό που κάνουν είναι να βοηθούν, για παράδειγμα, εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης να αποφασίσουν ποια έργα θα εντάξουν στα ΣΔΙΤ, στις συμπράξεις τομέα, για να είναι όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικοί. Δίνουν συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει καλύτερη λογοδοσία και δημόσια διαφάνεια. Επίσης, δίνουν συμβουλές έτσι ώστε να δομηθεί ένα έργο καλύτερα και να είναι περισσότερο επιλέξιμο και για άλλες επενδύσεις. Βοηθούν στην εξέβρεση χρηματοδοτικών ευκαιριών. Συμβουλεύουν για το πώς μπορεί κανείς να συνδυάσει το ΕΦΣΙ με το ΕΣΥΦ, πώς να αξιοποιήσει τα διαρθρωτικά ταμεία και το καθεξής. Άρα είναι μεγάλη ζήτηση για αυτές τις δράσεις, πράγματι. Μπορούμε όμως να βελτιώσουμε αυτή την υπηρεσία και το προσπαθούμε. Προσπαθούμε να το πράξουμε λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους τα διάφορα κράτη-μέλη. Αλλά και τα διά, τις διάφορες ανάγκες που να ανταποκρίνονται στα ε, συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα. Η συνάδελφος Επίτροπος Κρέτσου μπορεί να σας δώσει περισσότερες εξηγήσεις για το τι μέλη γενέστε με τα διορθωτικά ταμεία. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω όμως ότι δεν θα αφαιρεθούν κονδύλια από τις περιφέρειες. Ούτε τίποτα το ενδιαφέρον θα συμβεί με τα διαρθρωτικά ταμεία από πλευράς ε, χρημάτων και τρόπου αξιοποίησης και χρήσης αυτών των χρημάτων. Είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε τι μπορούμε να αλλάξουμε, τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουν τα πάντα και μάλιστα ταχαίως. Αυτός είναι ο τρόπος να εκφράσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. όχι μόνο βοηθώντας τους ανθρώπους να ζουν την καθημερινότητά τους, αλλά ενισχύοντας τις επενδύσεις για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και οι εργασιακές συνθήκες, για παράδειγμα, στις εξόγως απόκεντρες περιφέρειες. Την προηγούμενη εβδομάδα ή την προπροηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις ιδιαίτερες ευκαιρίες της εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Καταλαβαίνω πολύ καλά την κατάσταση. Πρέπει όμως να έχουμε ανοιχτό πνεύμα όταν αποφασίζουμε τη μεταρρύθμιση για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Άλλωστε η χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να προέλθει από ε, τραπεζικές δομές που βρίσκονται στην ενδοχώρα. Δεν χρειάζεται ξεχωριστή ε, σύμβαση ή συμφωνία με το τοπικό υποκατάστημα, ε, το τραπεζικό. Μπορεί να έρθει χρηματοδότηση μέσω των ε, τραπεζών που εδρεύουν στην ενδοχώρα και όχι στην εξόχως απόκεντρη περιφέρεια. Ξέρω ότι η Επίτροπος Κρέτσου ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Ε, ιδιαίτερο μέλημά μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το, η παρατήρησή σας, κυρία Σπυράκη, είναι πολύ ε, σωστή. Πράγματι, υπάρχει βούληση να υπάρξει βοήθεια και να βοηθήσει κάποιος θέλει και να λάβει τη βοήθεια κάποιος άλλος θέλει. Ε, ε, ε, παρεμβαίνει όμως μια διαδικασία δυσχερής που καθιστά ανέφικτη ενδεχομένως την παροχή αυτής της βοήθειας ή και τη λήψη αυτής και αυτό είναι πραγματικά ματαιωτικό θα έλεγα. Ίσως πρέπει να εκπαιδευτούν καλύτερα οι άνθρωποι για τα μέσα, για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν καλύτερα αυτά τα μέσα. Σε κάθε περίπτωση το ΕΦΣΥ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, μπορεί να στηρίξει και πολύ μεγάλα έργα αλλά και πολύ μικρά. Και όταν γίνεται λόγος για μικρότερα έργα, ουσιαστικά μιλούμε για ε, χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που εντάσσονται στο δίκτυο μεσαίας κεφαλαιοποίησης. «20 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να είναι η αξία, η αξία κάθε έργου για να είναι επιλέξιμο στο ΕΦΣΥ. Βέβαια δεν υπάρχει κανένας νόμος που να απαγορεύει να είναι μικρότερη η αξία, όμως επειδή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν έχει τέτοιου είδου κατόφλι, πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί ε, η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να είναι και σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα, δηλαδή πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμα. Τώρα, 90.000 ευρώ είναι το χαμηλότερο έργο που άκουσα, η, αξία του, η χαμηλότερη αξία για έργο που άκουσα ότι έχει ε, ε υποβληθεί έτοιμα για χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτού του έργου. Στην Ελλάδα έχουμε δύο έργα και είμαι πολύ ικανοποιημένο για αυτά. Το ένα σε μια βιομηχανική περιοχή στον τομέα της μεταποίησης τροφίμων και το άλλο έργο έχει να κάνει με, ένα, με μια μικρομεσαία επιχείρηση. Υπάρχει μια συμφωνία και θα υπάρξει χρηματοδότηση ε, σε Έλληνες επιχειρηματίες ε, μέσα από μια συγκεκριμένη πλατφόρμα η οποία είναι επιλέξιμη για τη βοήθεια και θα διοχετεύσει τη βοήθεια σε Έλληνες επιχειρηματίες. Όλα αυτά ε, είναι στοιχεία που μας ικανοποιούν. Τα αποτελέσματα πείθουν. Πρέπει όμως να ε, κάνουμε ευαισθητοποίηση, να ε, ε, διαδώσουμε περισσότερο αυτό το μήνυμα. Από την προηγούμενη μου εμπειρία εκτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαθαίνω ότι όταν πια έχεις ήδη στείλει το μήνυμά σου χιλιάδες φορές τόσο που δεν αντέχεις πια να το επαναλαμβάνεις, τότε είναι που ίσως πραγματικά έχει φτάσει σε όλα τα αυτιά που πρέπει να φτάσει. Επομένως, ας συνεχίσουμε ε, να ε, αναμασούμε τα ίδια και τα ίδια, προκειμένου να διαδώσουμε όσο το περισσότερο αυτό το μήνυμα. Ε, μπορούμε να βρούμε αυτές τις ε, πληροφορίες στο site, αλλά ε, πότε θα έχουμε την ενδιάμεση αξιολόγηση τον Ιούνιο, οπότε πότε, πιανού χρόνου, τον Ιούνιο πιανού χρόνου. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αξιολογεί το ΕΦΣΙ σε τακτική βάση. Και νομίζω ότι η αξιολόγησή της θα είναι έτοιμη τον Ιούνιο είναι η τακτική έκθεση τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το μέλλον του ΕΦΣΥ προβλέπεται να ελεγχθεί και να εξεταστεί ξανά το Μάρτιο του επόμενου έτου, σύμφωνα με την νομοθεσία. Θα εξετάσουμε τις αδυναμίες και τα ατού του ΕΦΣΥ και να δούμε, για να δούμε αν πρέπει να αλλάξουμε τον κανονισμό του. Ο ίδιος ο κανονισμός προβλέπει ότι η αξιολόγηση της συνέχισης του ΕΦΣΥ θα πρέπει να γίνει μέχρι το Μάρτιο του 2017. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Κατάινεν. Ήταν πολύ χρήσιμη και ωφέλιμη αυτή η συζήτηση και ελπίζω δεν ήταν η τελευταία μας συνάντηση. Είστε καλοδεχούμενοι. Okay, uh, Ας κλείσουμε τη σημερινή συνεδρίαση. Επόμενο σημείο, τα διάφορα. Έχουμε κάτι στα διάφορα. Όχι. Επόμενη συνεδρίαση, σας υπενθυμίζω ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι ήδη αύριο. Έκτακτη συνεδρίαση από τις 7 μετά μεσημβρία. Ανταλλαγή με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ντομπρόφσκης. Κλείνουμε το δημόσιο κομμάτι της συνεδρίασής μας και θα συνεχίσουμε και κλεισμένο το θυρών με τις συνεδρίες των συντονιστών. Ευχαριστώ πολύ τους διερμηνείς. Εκ μέρους όλων. Ευχαριστούμε.